Ladies Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ και καλησπέρα σας. Let me restart the... Ας αρχίσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθως, αλλά το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, όσο και ενδιαφέρον. Έχουμε μια δημόσια ακρόαση με θέμα τη διάσταση της ασφάλειας της αλλαγής του κλίματος. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, ερωτηματικό, για την Ευρω... κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Έχουμε τέσσερα διακεκριμένα μέλη του πάνελ. Ε, θα ήθελα να τους ε, καλωσορίσω. Είναι ο κύριος Ντομινίκ Πόρτερ, ε, ε ασχολείται στην υπηρεσία εξωτικής δράσης με παγκόσμια θέματα και οικονομικά. εδώ εξεβωνήμων. Έχουμε τον κύριο Λούκας Ρίτιγκερ, ο οποίος ε, είναι ανώτερος τέλεχος διαχείρισης προγραμμάτων ε, στο Adelphi Research και επιπλέον του ανατέθηκε η μελέτη για το ίδιο θέμα ε, της κλιματικής αλλαγής. από την ομάδα των 7. Κατέθεσα τη μελέτη στο G7. Ελπίζω να ακούσουμε για αργότερα μερικά σχόλια. Σταματώ εδώ σχετικά. Εδώ στα δεξιά μου, μετά τη γραμματεία, είναι ο καθηγητής Τόρ Μπενιαμίνσεν, ε, καθηγητής ε, από την Νορβηγία, πανεπιστημιακός, ε, στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Βιολογικών Επιστημών, στο ε, Πανεπιστήμιο της πόλης ΟΣ στην Νορβηγία και θα μας ενημερώσει για θέματα κλιματικής αλλαγής και ασφάλειας. Not least as Και τέλος, χωρίς καθόλου να είναι λιγότερο σημαντική παρουσία, η πρόσωπος ενός think tank και ηγετικού Ινστιτούτου ε, έχουμε συνεργασία με την υποεπιτροπή μας γιατί μας παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη, πράγματα γνωμοσύνη και την ευχαριστούμε. Είναι η κυρία Μάλιν ε, Μόμπιορκ, ανώτερη ερευνήτρια στο ΣΥΠΡΙ, το οποίο είναι το Κέντρο Διεθνούς Έρευνας για την Ειρηνή στη Στοκχόλμη. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ντόμινικ Πόρτερ. Παρακαλώ. Thank you very much indeed uh, for the introduction. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκλησή σας σήμερα, να παραστώ εδώ σήμερα στην υποεπιτροπή σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα κάνουμε νομίζω όλοι ό,τι μπορούμε όχι μόνο να δείξουμε ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα, αλλά θα προσπαθήσουμε να το καταστήσουμε και ενδιαφέρον, όπως είπατε και εσείς. Εγώ μιλώ για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ε, ασφάλειας, κλιματικής ε, ασφάλειας. Θα προσπαθήσω εισαγωγικά να κάνω μία παρουσίαση του θέματος, να προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί είναι σημαντικό και οι προηγούμενες προσπάθειές μας, ε, τι ακριβώς ήταν και τι ακριβώς κάνουμε ε, και πώς ε, σχετίζονται με το θέμα. Ξεκινάμε με μια πεποίθηση για τη σύνδεση μεταξύ της ασφάλειας και της κλιματικής ασφάλειας. Θα σας πω ένα πράγματα για το αφεντικό μου. Η Φεντερίκα Μοντερίνη κάνει αυτή την σύνδεση συνεχώς στην ε, διάσκεψη ασφαλείας στο Μόναχο είπε φέτος ότι όταν επενδύει κανείς στην ανάπτυξη, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, επενδύεις και στην δική σου ασφάλεια. Απλό είναι αυτό νομίζω και κατανοητό. Η επίσημή μας θέση ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, στην οποία κατέληξαν το Μάρτιο του τρέχοντος έτους τα κράτη-μέλη. Θα σας πω λοιπόν τα συμπεράσματα ε, του G7 και του G20 ε, σε διάφορα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς ότι πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση των κλιματικών αλλαγών με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα ε, να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα, να προβλέψουμε και καλύτερα ε, τη σημασία της κλιματικής αλλαγής όσον αφορά την ασφάλεια και την μετατόπιση των πληθυσμών. Αυτή λοιπόν είναι η επίσημη γραμμή μας, η επίσημη άποψη του τι πρέπει να κάνουμε. Φυσικά τα λόγια δεν είναι αρκετά. Θα ήθελα να πω όμως ότι το να το συζητούμε, να μιλάμε γι' αυτό είναι σημαντικό από μόνο του η κλιματική διπλωματία είναι κάτι που μας επιτρέπει να προσθέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ορατότητα στους υπέρμαχους ε, ε, του κλίματος σε διάφορες οικονομίες, ώστε οι οικονομολόγοι να συμμετέχουν και εκείνοι στην προσπάθεια, οι ενεργειακές ε, εταιρείες, οι όσοι ασχολούνται με τα θέματα ασφαλείας, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι το ο ε, οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουν το βάρος της ε, σημασίας της πολιτικής τους. Ε, υπάρχει ας πούμε η παραδοσιακή περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική μπορεί κατά κάποιο τρόπο να παραγωνίζεται από την επίσημη πολιτική ηγεσία σε τέτοια θέματα. Οπότε αυτό θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσουμε από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ε, σύνδεση είναι όλα αυτά να ε, ενταχθούν ε, στις δράσεις διαχείρισης κρίσεων ή το να τις σχεδιάζουμε ή όταν πρέπει ήδη να περάσουμε στην πράξη αντιμετώπιση κρίσεων, αντιμετώπιση περιβαλλοντικών καταστροφών, αναπτυξιακή πολιτική, ο συνδυασμός όλων αυτών των πτυχών νομίζω ότι εντάσσεται ε, σωστά ε, στην εξωτερική ε, πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρώτον πρέπει να εντοπίσουμε ποια είναι η πτυχή ασφαλείας της κλιματικής αλλαγής, ε, σε τι μορφές εκδηλώνεται, για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Θα ήταν πολύ απλοϊκό να πούμε ότι όλοι οι παράγοντες πίεσης η περιβαλλοντική σε μία ε, σύγκρουση, για παράδειγμα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είπε προσφάτως ότι 40% των ένοπλων ε, συγκρούσεων του τελευταίου αιώνα συνδέθηκαν με, συνδέονται με περιβαλλοντική παράγοντε. παράγοντες, ε, αλλά τώρα κατά πόσο αυτό συνδέεται στη συνέχεια με κλιματική αλλαγή είναι δύσκολο να το καταδείξουμε αυτό. Μερικέ φορέ ε, υπάρχει υπερβολική εκμετάλλευση ή εξάντληση των ε, φυσικών πόρων που είναι το αποτέλεσμα μια ένοπλη σύραξη. Αυτό ισχύει από καταβολή κόσμου, δεν είναι κάτι το καινούριο. Ε, Προφανώ ο κόσμο πάντοτε πολεμούσε για πολύ περιορισμένου πόρου. Ε, οι συνάδελφοι μπορεί να το γνωρίζουν πολύ περισσότερο. Ε, η κλιματική αλλαγή λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής της απειλής. Είναι ένας παράγων ο οποίος ε, ε, φορτώνει περισσότερο τις υπάρχουσες πιέσεις και αυξάνει τις πιθανότητες αστάθειας και βίαιων συγκρούσεων. Λοιπόν, είναι ένας παράγων ο οποίο ε, συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Ε, για παράδειγμα υπάρχει καταστροφή εσοδίας ε, υπάρχουν λιγότερα τρόφιμα, υπάρχουν υψηλότερες τιμές, μειώνεται η ασφάλεια των οικοκυριών υπάρχει εξαναγκαστική μετανάστευση, υπάρχει έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα, σε πλημμύρες, σε κατακλυσμούς, υπάρχει αύξηση της στάθμης της θάλασσας ε, που μπορεί να ε, ε, απειλήσει ειδικότερα παράκτιες περιοχές. Μπορώ να πω και άλλα παραδείγματα, αλλά οι παράγοντες συνήθως δεν είναι απομονωμένοι, συνήθως συνδέονται μεταξύ τους στο πλαίσιο του γενικότερου αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, ο αντίκτυπος που προέρχεται από το κλίμα και όλες οι πτυχές της που υπάρχει περίπτωση να φτάσουν σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο και να γίνουν μοιραίες, ε, ε, απλώς ε, προστίθενται στα ήδη, στη ήδη βεβαρημένη κατάσταση που υπάρχει διότι όσο λιγότερο ανθεκτική είναι μια ε, κοινωνία τόσο, ε, ε, και όσο επηρεάζεται από την κλιματική αλληλεγγύη, τόσο αυτοί οι παράγοντες που ανέφερα μπορούν να κάνουν τη διαφορά από κάτι που είναι σχετικώς διαχειρίσιμο σε κάτι το οποίο μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Να σας δώσω και μερικά παραδείγματα τώρα, πέρα από τη θεωρία ε, και υπάρχουν παραδείγματα που θα δώσουν οι συνάδελφοι από τον πραγματικό κόσμο, τα γνωρίζουν καλύτερα από μένα, αλλά καταστάσεις ε, πολύ ε, ανησυχητικές που μπορούμε να τα δούμε από αυτή την οπτική γωνία του κλίματος, όταν θεωρούμε δηλαδή ότι υπάρχει μια προληπτική δράση η οποία θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο. Να αρχίσω με τον κόλπο της Βεγγάλης, ένα πολύ μεγάλο, ε, ένα πολύ μεγάλη, μια πολύ μεγάλη περιοχή, Μπαγκλαντές, Μιανμάρ, βλέπουμε πολύ σημαντικές αλλαγές ε, στην, ε, κλιματική, στο κλίμα εκεί. Υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια, επηρεάζεται πολύ περισσότερο κόσμος, ε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, τα ανάντι του ποταμού, στην Κίνα για παράδειγμα, ε, στα Ιμαλάια οι χώρες αυτές πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και όχι να ανταγωνίζονται. Ε, εμένα μου φαίνεται λογικό αυτό. Η Αραβική Άνοιξη, να μιλήσουμε λίγο και για την Συρία και την απειλή ε, που έχει, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που είπα προηγουμένω, αύξηση ε, των τιμών ε, ε, των, τροφίμων λόγω της εξηρασίας, μία ανώτατη τιμή την οποία δεν μπορούσε η οποία ήταν πραγματικά κάτι που δεν, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί κανένας. Η, το, το τσάντ, για παράδειγμα, πολύ συχνά Η λίμνη του Τσάντ ε, είχε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Ε, έχει να αντιμετωπίσει πιο παρατεταμένες ξηρασίες ε, και αυτό βέβαια δημιουργεί πρόβλημα μεταξύ των αλλιέων, των βοσκών, ε, των γεωργών και των νέων που πολλούν πολύ δύσκολα να ε, ζήσουν από τις περιοχές, στις περιοχές στις ζούσαν. Ε, και έτσι αυτό αυξάνει και τον κίνδυνο εκμετάλλευση από ε, ομάδες όπως ε, η Αλσαμπάμπ και το Μποκοχαράμ. Ο κίνδυνο υπάρχει όχι μόνο στις φτωχότερε χώρε όμως. Θα ήθελα να το πω αυτό και θα ήθελα να αναφερθώ και στον ακτικό κύκλο. Όπως σας είπα, ε, λιώνουν οι πάγοι εκεί ε, και πέρα από όλες τις υπόλοιπες απειλές που σημαίνει αυτό για την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, υπάρχουν και μειότερα ε, μεταλλεύματα. Το πετρέλαιο και το αέριο δεν μπορούμε πια να τα εξορίξουμε. Ε, είναι ε, ένας, ένας κύκλος ο οποίος δεν είναι πια πάρα πολύ ε, υγιής από οικολογικής απόψεως και είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε. Ο κίνδυνος Βλέπουμε για παράδειγμα τις, τους κυκλώνες στην Λόνες ε, στην Καραϊβική που είχαν καταστροφικά αποτελέσματα, ε, χάθηκαν ολόκληρα ε, νησιά. Ήταν και, σε αυτή την περίπτωση όμως ο βαθμός προετοιμασίας, πρόληψης ε, και η ανθεκτικότητα της ε, πληγής σας κοινότητας έχει άμεση σχέση με το βαθμό και τη σοβαρότητα του αντικτύπου ε, στους ανθρώπους και στις υποδομές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν βλέπει κανείς τις ειδήσει, ακούει τις, τις εκθέσεις, τις ε, αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, από τους ε, από τις, για, την κατάσταση, το πώς οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ο τυφώνας αν θυμάστε καλά, το 2005 πέρασε από την Κεντρική Αμερική ε, σκότωσε πάνω από 10.000 άτομα στο διάβα του. Ε, αυτή τη φορά πήρε ίσως ένα διαφορετικό δρόμο ε, πάνω από πολύ πιο ευάλωτε περιοχές, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι ο αντίκτυπο ποικίλει ανάλογα με το που ζει κανείς και ακόμη και τότε ε, η κοινωνική αναταραχή που μπορεί να υπάρξει, το είδαμε μετά από τον τυφώνα Κατρίνα στι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι μια πολύ πλούσια χώρα, τα πράγματα μπορεί να ε, δυσκολέψουν, να οξυνθούν τα πνεύματα να ε, προχωρήσω τώρα στο τι κάνουμε εμείς, πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη αυτούς τους ε, παράγοντες ε, στο πλαίσιο των πολιτικών μας και πώς μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε πράξη. Όπως είπατε, τα παραδείγματα δείχνουν ότι είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, διαφορετικοί παράγοντες, διαφορετικός αντίκτυπος και για αυτούς τους λόγους πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ή τουλάχιστον μια πολύπλευρη ε, προσέγγιση με καλύτερη ε, προληπτική δράση. αύξηση της ευαισθητοποίησης είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, η διαχείριση του αντικτύπου μέσω μέτρων προσαρμογής επίσης. Αυτό νομίζω ότι είναι η κλασική δουλειά των ε, ε, αναπτυξιακών συστημάτων. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε πάρα πολύ καιρό. Μια διαδικασία διαλόγου με διάφορα μέρη του κόσμου, μακροχρόνια επενδυτικά προγράμματα που ελπίζουμε ότι στις πιο ευάλωτες περιοχές θα έχει αποτέλεσμα, θα υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις. Έχουν γίνει πολλά ακόμη και πριν ε, ε, να είναι απολύτως αναγκαία. Το 20% των δραστηριοτήτων μας έχει να κάνει έχουν να κάνουν ε, με την αντιμετώπιση, με τη διαχείριση των ποταμών και προσπαθούμε να δούμε με ποια μέτρα μπορούμε να με ποια προσαρμοστικά μέτρα μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όταν δούλευα στη Γενέβη, το, τη Οργάνωση, το ICRC, είδα ε, πώς έγινε η προετοιμασία για κάποιες κρίσεις. Ε, ήμουν με τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού. Ε, υπήρξε ένα κέντρο συντονισμού για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανταπόκριση στην κρίση. Ε, ήταν κάποιος, ε, ας πούμε, ένας συντονιστής που προσπάθησε να συγκεντρώσει ε, την ανάπτυξη όλων των μέσων και στρατιωτικών για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καταστροφές. Τώρα, συγκεκριμένα για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, αρχίζουν επιτέλους να ε, γίνονται συζητήσεις την περασμένη εβδομάδα, ε, την περασμένο μήνα συγγνώμη, από την ΕΙΕΔ, ε, θα σας πει και ο συνάδελφος περισσότερα, ήρθαμε σε επαφή με την στρατιωτική κοινότητα των κρατών μελών για να ακούσουμε και τη δική τους άποψη, τη δική τους αξιολόγηση για τον κίνδυνο που υπάρχει λόγω της αλλαγής του κλίματος. Υπάρχει επίσης και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο μας ε, ε, ε, βοηθά πολύ μας βοηθά να συμπεριλαμβάνουμε περισσότερο τους κινδύνους. Ε, είναι κάτι το οποίο το συμπεριλαμβάνουμε εγκαρσίως στις ε, πολιτικές μας, ε, με πολύ λεπτομερή τεχνική επιστημονική δουλειά, την οποία μεταξύ άλλων το Κοινό Κέντρο Ερευνών εκπονεί, μέχρι την αξιολόγηση του κινδύνου συγκρούσεων σε χώρες, οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι πιο ευάλωτες, επιλέγονται, βλέπουμε τις αντιπροσωπείες που υπάρχουν εκεί, οι ε, πρεσβείες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συζητούν, συντονίζονται για να δουν τι μπορούν να κάνουν για να υπάρξει μια πρόληψη ενδεχόμενης ε, κρίσης. Βέβαια χρησιμοποιούμε και επιστημονικά δεδομένα στο σχεδιασμό της πολιτικής μας. Βλέπετε ότι συντονίζουμε τις προσπάθειές μας και ελπίζουμε ότι αυτό αρχίσει σιγά σιγά να καρποφορεί. Ε, το greening, το πρασίνισμα ας πούμε της, ε, ε, των στρατιωτικών δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν τώρα ένα εγχειρίδιο όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία και την οικολογική αποτελεσματικότητα. Θέλουμε δηλαδή το αποτύπωμά μας άνθρακα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο όταν είμαστε όταν δραστηριοποιούμεθα σε ένα συγκεκριμένο ε, μέτωπο, προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα νέο μοντέλο ε, περιβαλλοντικής πολιτικής, πάντοτε σε συνδυασμό με ε, τη διοίκηση των στρατιωτικών μας δυνάμεων, αλλά όλα αυτά μου πάνε πίσω σε αυτό που ήθελα να πω στην αρχή, ε, ότι η ευαισθητοποίηση είναι πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι μπορεί ακόμη και οι στρατιωτικές δυνάμεις να μας βοηθήσουν στο να το επικοινωνήσουμε αυτό καλύτερα και πέρα από τη δική τους ε, πολύ περισσότερο ε, από ό,τι θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια πιο αισιόδοξη νότα, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι εύκολο στο ε, θέμα αυτό που πραγματεύομαι. Ε, Πιέζουμε για συνεργασία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μεταξύ των κρατών, στο πλαίσιο των οργανισμών ε, και από τους οργανισμούς για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές για την ασφάλεια που προέρχονται από το κλίμα. Η δική μου αίσθηση είναι ότι θα μπορούσε να υπάρχει ε, ένα διπλό αποτέλεσμα αν οι ενδιαφερόμενοι φορείς αυτών των hot spots ε, να συγκεντρωθούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να βοηθήσουν την κατάσταση. Ε, βέβαια, πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρωτοστατούν στην προσπάθεια ύπαρξης πιέσεων ώστε να γίνει κάτι τέτοιο και η Σουηδία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο φέτος και του χρόνου με τους εταίρους μας όλο τον κόσμο αλλά ακόμη και σε δίκτυα σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο πόλεων που μπορεί να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Προσπαθούμε να συνεργάζονται, να συνομιλούν για να μπορούν να εντοπίζουν καλύτερα κοινέ προσεγγίσεις ή τουλάχιστον να ανταλλάσσουν εμπειρίε. Να συνεργάζονται δηλαδή οι άνθρωποι πριν ο αντίκτυπο του, της κλιματικής αλλαγής τους χωρίσει. Ε, επειδή το είπε αυτό ο Πρωθυπουργό ε, των Φίτζη στη Βόνη την περασμένη εβδομάδα, είμαστε όλοι στο ίδιο κανό, είπε. Ε, και είναι η δουλειά μας να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το κανό ε, θα φτάσει ε, με ασφάλεια στον προορισμό του. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ κάνω, κάνω και ξέρω ότι είναι ένα μικρό σκάφος. Οπότε είναι δύσκολο να είναι κανείς μαζί με άλλους πάνω στο κανό. Ο ε, Λούκας Ρίτιγκερ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την εισαγωγή. Εγώ θα πω κάποια πράγματα σε σχέση με τις ενδείξεις ασφάλειας της κλιματικής αλλαγής για την Ένωση και θα επικεντρωθώ σε κάποια ζητήματα που αναφέρθηκαν όσον αφορά τις πολιτικές, τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή για τους κινδύνους κλπ. Ξεκινώντας να πω ότι τα τελευταία 10 με 15 χρόνια η γνώση μας για την σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής και ασφαλείας έχει αυξηθεί σημαντικά. Και αυτό φαίνεται, φάνηκε το 2014, όπου για πρώτη φορά είχαμε μια έκθεση για το κλίμα με ένα κεφάλαιο για την ανθρώπινη ασφάλεια η οποία απειλείται λόγω κλιματικής αλλαγής και επίσης είχαμε διάφορες εκθέσεις και μελέτες για το θέμα. Ήδη η, ο στρατός στην Αμερική άρχισε να το εξετάζει το θέμα και το 2007 είχαμε ένα κέντρο ανάλυσης που είχε αυτή την έκθεση σε σχέση με την απειλή δηλαδή που παρουσιάζει η κλιματική αλλαγή όσον αφορά τα τροτικά θέματα. Το 2015 είχαμε μια έκθεση από το G7 που μας είχαν αναθέσει για να μιλήσουμε αυτό το θέμα και να χαράξουμε συστάσεις και τευθυντές γραμμές γιατί μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου. Επίσης, Κατά διάρκεια της παρουσίασής μου θα σας παρουσιάσω κάποια από τα ευρήματά μας στην ανάλυση αυτού του κινδύνου και κάποια συγκεκριμένα ευρήματα όσον αφορά την σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής, τρομοκρατία και μετά θα αναφερθώ και σε συστάσεις, τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή. Ως πήμα λοιπόν της ανάλυσης κινδύνου του νέου κλίματος για την ειρήνη, εμείς εξετάσαμε το πώς επηρεάζονται οι συνθήκες ασφαλής από την ε, κλιματική αλλαγή και τι παραγόντες υπάρχουν. Είδαμε ότι δεν υπάρχει μια απλή σχέση γενεσιουργός δηλαδή μεταξύ κλίματος και σειράξεων. Όμως είδαμε επίσης και αυτό ήδη αναφέρθηκε και προηγουμένως ότι η κλιματική αλλαγή συγκλίνει με άλλες πιέσεις και αυτό οθεί τις κοινωνίες προς κάποια ευαισθησία, κάποια αδυναμία, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ε, κλιμάκωση βεβαίως σειράξεων και βίας. Δηλαδή έχουμε ένα πολλαπλασιαστή κινδύνου την κλιματική αλλαγή. Αυξάνεται λοιπόν η πίεση όσο αυξάνεται η κλιματική αλλαγή, συγκλίνει με άλλες μεγάλες τάσεις όπως η αύξηση του πληθυσμού, η αύξηση τη αστικοποίηση, η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Έχουμε 7 κινδύνους αδυναμίας που απορρέουν από, το, από την κλιματική αλλογή. Θα του αναφέρω και θα αναφέρω και δύο παραδείγματα. Ο πρώτος κίνδυνο είναι οι σειράξεις για τοπικούς πόρους επειδή ακριβώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους φυσικούς πόρους όπως ε, το έδαφος και τα ύδατα. Υπάρχει έλλειψη, υπάρχει σπάνη. Οπότε υπάρχουν πιέσεις και υπό κάποιες συνθήκες ή προϋποθέσεις υπάρχει μια δυναμία που οδηγεί σε, ενδεχομένως σε συγκρούσεις. Αυτές οι συγκρούσεις μπορούν μετά να κλιμακωθούν. Ή αυτός ο ανταγωνισμός μπορεί να κλιμακωθεί και να οδηγήσει σε συγκρούσεις και βία. υπό διάφορε μορφέ που θα αναφέρουν και οι συναδελφοί στη συνέχεια. Σήμερα έχουμε σειράξει γύρω από πόρου που αφορούν τι εξορίξει. Κάτι το οποίο έχει και με, όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν πολλαπλασιάζει αυτές τις δυναμικές κινδύνου και αναμένουμε να αυξηθούν μελλοντικά. Ο δεύτερος κίνδυνος αδυναμίας είναι η ασφάλεια του ανθρώπινου πληθυσμού και μετανάστευση. Βέβαια, λόγω ελλείψης πόρων όπως νερό κτλ. Πολλές ομάδες πληθυσμού εξαρτώνται άμεσα από αυτούς τους πόρους, ας πούμε πολύ εξαρτώνται από την γεωργία, οπότε αυτή η ανασφάλεια του πληθυσμού τους οδηγεί στο να ομαδοποιούνται, να αναζητούν εναλλακτικέ λύσεις υπό μορφή ας πούμε, παρανόμων δραστηριοτήτων, παραγωγή ναρκωτικών ας πούμε, στο Αφγανιστάν και αλλού, ή μπορεί να δημιουργήσει ή να αποτελέσει μια όθηση για τη μετανάστευση, όπως ξέρουμε σήμερα. Να πω παράλληλα ότι αν δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή και πώς αναμένουμε να εξελιχθούν αυτές οι κινήσεις, βλέπουμε ότι αυτές οι μετακινήσεις συμβαίνουν εντός των χωρών δηλαδή από τις αγροτικές περιοχές στις πόλεις. Και σε πολύ ακραίες περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν μακροχρόνιες ή μεγαλύτερες κινήσεις εντός ας πούμε υπήρων ή όπως τώρα με την σύγκρουση στην Συρία όπου ένα μικρό τμήμα αυτού του πληθυσμού έφτασε εδώ στην Ευρώπη. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι θεομηνίες αναφέρθηκαν σήμερα και η υποβάθμιση της ασφάλειας είναι σημαντικό γεγονός μετά από θεομηνίες. Οπότε το κράτος θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει ασφάλεια, αλλά κυρίως να μπορέσει να επαναφέρει την ασφάλεια και πόρους όπως τα ύδατα. Όλα αυτά σχετίζονται με την ανταπόκριση της κυβέρνησης στις θεομηνίες, ιδιαίτερα όταν αυτές οι θεομηνίες είναι πολλαπλές. Θα πρέπει να δούμε ετησίως πώς αντιδρούν οι κυβερνήσεις και πώς προσλαμβάνουν την ένταση αυτή οι πληθυσμοί. Αν φτάνει ή δεν φτάνει, αυτό οδηγεί βεβαίω σε αμφισβητήσει τη κυβέρνηση και υπάρχουν και πολλά πρακτικά παραδείγματα γι' αυτό. Επίση, σήμερα αναφέρθηκε ένα θέμα που έχει ερευνηθεί, δηλαδή πολιτική αστάθεια και η ταχεία αύξηση τη τιμή των τροφίμων. Το 2011, α πούμε, είδαμε ότι οι τιμέ των τροφίμων αυξήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα παγκοσμίω και αυτό οδήγησε καταλητικά σε πολιτική αστάθεια σε διάφορες χώρες. Αίγυπτο, Αραβική Άνοιξη, η αύξηση ας πούμε του Άρτου ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας στις ταραχές εκεί. Διαχείριση υδάτων. Και αυτό αναφέρθηκε σήμερα. Εδώ δεν έχουμε πολλά παραδείγματα από το παρελθόν όπου η σειράξει για το νερό, οι διασυνοριακέ οδηγούν σε βίε σειράξει ή συγκρούσει. Μα απασχολεί όμω, μα ανησυχεί το ερώτημα αν η υπάρχουσα διαχείριση υδατίνων πόρων στον Ήλο, στην Ινδία και αλλού, αν Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή αντιμετώπιση από την συνεχόμενη και αυξανόμενη πίεση του πληθυσμού και τη περιβαλ... κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μα απασχολεί ιδιαίτερα και το παρελθόν θα πρέπει να μα καθοδηγήσει για το μέλλον. Αύξηση του... τη στάθμη τη θάλασσα βεβαίω. Είναι υπαρξιακή αυτή η απειλή για κάποια μικρά νησιά, αλλά πρέπει να πούμε ότι ήδη η αύξηση τη στάθμη τη θάλασσα έχει αντίκτυπο ήδη από τώρα. Έχουμε δηλαδή καταιγίδε και αύξηση του κινδύνου ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Μπαγκλαντές ή ο κόλπος Βενγκάλης που αναφέρθηκε προηγουμένως, όπου αυτοί οι κίνδυνοι ήδη υπάρχουν σήμερα. Ο τελευταίος κίνδυνος από την κλιματική αλλαγή είναι κάπως διαφορετικός. Εμείς ε, εξετάσαμε, δεν εξετάσαμε μόνο δηλαδή, την ανταποκρισή μας, αλλά πολιτικές μετρίασεις και τις ανεπιθύμητες αρνητικές ενέργειες που μπορεί να έχουν. Επειδή αυτές οι πολιτικές είναι πια ευρείες και όπως οποιαδήποτε άλλη πολιτική μπορούν και αυτές να έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε με πλαίσια αδυναμίας και συγκρούσεων, οπότε θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην αυξήσουμε τις δυναμικές σύγκρουσης. Βιοκαύσιμα, ένα άλλο ένα παράδειγμα του παρελθόντος, όπου οι πολιτικές μετρίασεις είχαν γιατί ε, ε, τα επιδόματα είχαν πολύ ευρείες επιπτώσεις που οδηγήσαν στην επέκταση των καλλιεργιών σε πολλά μέρη όπως η Νότια Αμερική και αυτό οδήγησε στην αποψήλωση και σε συγκρούσεις για τη γη. Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό να το έχουμε κατά νου σε σχέση με την εφαρμογή, δηλαδή την ευρεία πια εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Όπως υποσχέθηκα πριν, να δώσω και δύο παραδείγματα. Καταρχάς Συρία. Πριν από την σύγκρουση, το 2005 και το 2006-2011 είχαν τη χειρότερη χρονιά ξηρασίας. Και αυτό είχε φοβερές επιπτώσεις όσον αφορά την ζωή μεγάλων πληθυσμών, ιδιαίτερα των γεωργών στη βόρεια χώρα, όπου περίπου το 85% του ζωικού κεφαλαίου απεβίωσε και ένα εκατομμύριο αναγκάστηκαν να μετακινηθούν. Αυτό συνέβαλε στη μετακίνηση μεγάλου, κομμάτι, μεγάλου κομματιού πληθυσμού από την ύπεθρο της πόλεις. Υπάρχει πολύ, ε, πολύ ψηλό επίπεδο πληθυσμού, δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς ε, επίσης πρόσφυγες από το Ιράκ που πήγαν εκεί και το 2011 επίσης όταν είχαν πολύ ψηλέ τιμές τροφίμων όλα αυτά οδήγησαν σε μια ανθρωπιστική κρίση και αυτή η ανθρωπιστική κρίση συνέβαλε στο ξέσπασμα των ταραχών. Δεν θα ήθελα να πω ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί το μοναδικό παράγοντα ή είναι το μόνο που οδήγησε στην σύγκρουση στη Συρία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς αυτή η κλιματική αλλαγή ε, διαδρά με άλλες πιέσεις και είχαμε μια αυταρχική κυβέρνηση που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το αυξανόμενο αίτημα για δημοκρατία και ειρήνη πλημμύρες στην Ταϊλάνδη, το 2011 επίση. Είχαμε τις ε, μεγαλύτερες ε, βροχοπτώσεις ε, την τελευταία 30 ετία σε μεγάλο τμήμα της χώρας, σε μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση πολιτικά. Είχαμε μια νέα κυβέρνηση, η οποία μόλις είχε αναλάβει καθήκοντα και αυτή η θεομηνία ήταν μια δοκιμασία για την κυβέρνηση αυτή που σε σχέση με τον πληθυσμό που την ψήφισε και τις προσδοκίες του και πρέπει να πούμε ότι απογοήτευσε αυτό τον πληθυσμό. Οπότε ο πληθυσμός θεωρήσε ότι η παροχή βοήθειας δεν ήταν διαφανής, δεν ήταν δίκαιος και αυτό απαιτέλεσε μια καταλυτική ε, ένα καταλητικό παράγοντα για τις ε, ταραχές που είχαμε στη συνέχεια. Ένα τελευταίο σημείο για τους κινδύνους που θα ήθελα να το διευρύνω λίγο. Κλιματική αλλαγή και παραστατικές οργανώσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις και οργανωμένο έγκλημα. Εμείς γράψαμε μία έκθεση για αυτό το θέμα, για τη σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής και παρακρατικών οργανώσεων και είδαμε ότι δεν δημιουργεί τρομοκρατία κλιματίες Η κλιματική αλλαγή, αλλά συμβάλλει στη δημιουργία ενός ε, πλαίσιών περιβάλλοντος όπου μπορούν να ευδοκιμήσουν αυτές οι οργανώσεις. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να δράσουν πιο ελεύθερα. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν συνέβαλε στο να υπάρχει περισσότερη δυναμία και άνοιξε ένα παραθυράκι αυτές τις ομάδες. Οι ομάδες μάλιστα από ομάδες οι οποίες ανέλαβαν και ε, ρόλο εξουσίας, κράτους σε αυτές τις περιοχές. Και μάλιστα προσελκύουν νέους αυτές οι παρακρατικές οργανώσεις, ε, νέους οι οποίοι δεν έχουν καμιά προοπτική στη ζωή τους. Γιατί είναι λοιπόν σημαντικό σε αυτό το περικολό πλαίσιο να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση σε πολιτικό επίπεδο να Μιλάμε για, το, για τη τρομοκρατία και τις τρομοκρατικές ομάδες. Βλέπουμε όμως ότι η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Θα πρέπει να ευρύνουμε τις οριζοντές μας εδώ. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ακριβώς τα κίνητρα και το περιβάλλον μέσα στα οποία, μέσα στο οποίο ευδοκιμούν αυτές οι ομάδες. Μόνο τότε θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, απειλές και τους κινδύνους που παρουσιάζουν αυτές οι παρακρατικές οργανώσεις. Επανερχόμενος τώρα στους 7 κινδύνους αδυναμίας που ανέφερα προηγουμένως, μίλησα για περιπλοκότητα και περιπλοκότητα με αυτό εννοούμε τους κινδύνους που απορρέουν από την διάδραση αυτών των παραγόντων αλλά αυξάνουν, οξύνουν ο ένας παράγοντας το άλλο αυτό σημαίνει ότι έχουμε συστημικούς κινδύνους και αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους, αυτές τις ομάδες συστημικών κινδύνων θα πρέπει οι πολιτικές μας να περιλαμβάνουν αυτή την, ε, αυτό χαρακτήρα με πολλές διαστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενσωματώσουμε συγκεκριμένες πολιτικές σημαντικές πολιτικές αναφέρθηκε οπότε δεν επαρκεί πια να δουλεύουμε παράλληλα ή διαστρωματικά. Θα πρέπει να έχουμε συνολικότερε πολιτικέ, θα πρέπει να αναπτύξουμε βεβαίω τη συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και θα πρέπει να έχουμε και δραστηριότητε αποτροπή σειράξεων και ειρήνη και θα πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να δημιουργήσουμε γέφυρε σε όλε αυτέ τι θεμακέ πολιτικέ. Ο κύριο μα στόχο βέβαια παραμένει το να επικεντρωθούμε στην πρόληψη και στο να εστιάσουμε στην αντοχή κατά των κινδύνων ε, αδυναμίας που παρουσιάζει η κλιματική αλλαγή. Και να πω μάλιστα εδώ ότι η κλιματική αλλαγή ως απειλή δεν σημαίνει ότι εμείς θεωρούμε ότι οι απαντήσεις σε αυτούς τους κινδύνους σημαίνει περισσότερη αστυνόμευση. Οι περισσότεροι στρατιωτικοί και οι υπεύθυνοι των πληροφοριών συμφωνούν ότι ο στρατός η στρατικοποίηση δεν αποτελεί τη λύση. Βεβαίως διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο και συμμετέχει ενεργά ως συνιστό. Αυτό αφορά βέβαια και την εξωτερική πολιτική. Έχουμε την ε, ε, κλιματική διπλωματία και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης νομίζω ήταν πρωτοπόρος αυτό, στην κλιματική δηλαδή διπλωματία, στην στρατηγική που επικεντρώνεται στην κλιματική αλλαγή. Αυτό θα, θα πρέπει να συνεχιστεί. Όμως θα πρέπει να είμαστε σοβαρότεροι σε σχέση με το να πάμε πέρα ε, της διαχείρισης των κρίσεων στα πλαίσια της κλιματικής διπλωματίας. Αυτό είναι δύσκολο γιατί ήδη έχουμε περισσότερες κρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε δύσκολα. Θα πρέπει λοιπόν να μετατοπιστούμε από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες κρίσεις με προοπτικές δράσεις. οι λεκάνες απορροής. Εκεί υπάρχει μεγάλο πεδίο εντάσεων. Εκεί θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε αποτρεπτική δράση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως η εξωτερική πολιτική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την διασφάλιση συνοχής της πολιτικής. Οπότε αυτοί που χαράσουν αυτές τις πολιτικές είναι σε καλύτερη θέση για να ξέρουν ακριβώς πώς θα μπορούσε να κληρωθεί αυτή η ενσωμάτωση, να γίνει αυτή η ολοκλήρωση και στον τομέα επίση τη αποτροπή. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον αμοιβαίο διάλογο στο διεθνέ πλαίσιο. Θα πρέπει να ασφαλίσουμε το ότι η Συμφωνία των Παρισίων δεν θα πρέπει να εγκαταστήσει βέβαια την βοήθεια για την ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να, να εφάπτονται και να έχουμε και τα κατάλληλα συστήματα, όπω το σύστημα του ΟΗΕ. Εδώ διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι ανθρωπιστικέ οργανώσει, αλλά και η ανάπτυξη οι θεσμοί μάλλον ανάπτυξης όπως Παγκοσμία Τράπεζα ή δομές όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτοί που χαράσουν εξωτερική πολιτική λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτοί οι θεσμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους σοβαρά αυτούς τους κινδύνους και να παράσχουν απαντήσεις. Συνεργασία για την ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια. Και εδώ θα πρέπει να βελτιωθούμε όσον αφορά την πρόληψη. Νομίζω ότι Για κάθε ευρώ που δαπανούμε για την πρόληψη γλιτώνουμε 4 με 7 ευρώ όσον αφορά την ανταπόκρισή μας στην οικονομική και αυτό θα ξεκινήσει μέσω της ανάπτυξης της ανθρωπιστικής βοήθειας και της συνεργασίας για την ανάπτυξη και θα πρέπει να πάμε πέρα από τα συμπτώματα απλά και μόνο. Αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένω. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη, μεγάλο όγκο ανθρωπιστική βοήθεια πάει σε αυτήν την περιοχή. Όμω από μόνη τη ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα λύσει το πρόβλημα. Παρόλο λοιπόν που υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, μια από τι μεγαλύτερε στον κόσμο, ακόμα θα πρέπει να σκεφτούμε το πώ θα τα συνδέσουμε όλα αυτά με αυτό που συζητάμε, αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να τα λύσουμε. Ένα άλλο λόγο για τον οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε αυτέ τι διαστρωματικέ προσεγγίσει, είναι ότι έχουμε μορφές χρηματοδότησης οι οποίες είναι αποσπασματικές συνεργασία για την ανάπτυξη κτλ. Θα πρέπει όλα αυτά να είναι ολοκληρωμένα, ενσωματωμένα και να ακολουθούν την εφαρμογή προγραμμάτων που και αυτά θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα. Δηλαδή υπάρχουν καλά παραδείγματα από την Ευρώπη. Υπάρχουν εργαλεία την σταθερότητα και την ασφάλεια με κατάλληλα προγράμματα για την δημιουργία ειρήνης, για την ειρήνευση και αυτά είναι πολύ αποδοτηματικά είναι σημαντικά και τα χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα. Και με αυτό φτάνω στο τελευταίο μου σημείο για την διασύνθεση μεταξύ ειρήνευσης και κλιματικής αλλαγής. Έχουμε λοιπόν προγράμματα τα οποία αντιμετωπίζουν κλιματικούς κινδύνους και σειράξεις. Έχουμε χρηματοδότηση από την Ένωση ας πούμε, προγραμμάτων που θα επικεντρωθούμε στο Νεπάλ και το Σουδάν και τα προγράμματα που έχουμε εδώ αναπτύσσονται και θα πρέπει να διαχέονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ενσωμάτωσή τους. Δύο λόγια για περιβαλλοντική πολιτική. Βεβαίω, η, η μετρίαση είναι μια από τι κυριότερε πολιτικέ μα. Ο περιορισμό, α πούμε, τη θερμοκρασία είναι πολύ σημαντικό. Αν όμως είμαστε σε θέση να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε πετύχει, αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ε, τα επόμενα, τις επόμενες δεκαετίες. Το οποίο σημαίνει θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προσαρμογές, δηλαδή περισσότερη χρηματοδότηση, αλλά να, να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η χρηματοδότηση θα καταλήξει σε συνθήκες και σε περιβάλλοντα αδυναμίας. όπου θα έχουμε συνεράξεις. Γιατί εκεί υπάρχει μεγαλύτερη αδυναμία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι αν αρχίσουμε τις επενδύσεις σε αυτές τις χώρες, τα προγράμματα προσαρμογής θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλα αυτά που συζητάμε και εδώ θα πρέπει οι ειδικοί να μην είναι απομονωμένοι αλλά να συζητήσουν ας πούμε, αυτούς που ασχολούνται με την ειρήνευση. Αλλιώς δεν τρέχουμε τον κίνδυνο να αξίνουμε αυτές τις ε, περιοχές όπου ήδη υπάρχουν σειράξεις. Τέλος, δύο λόγια για την άμυνα και την πολιτική ασφάλεια. Ο στρατός παγκοσμίως έχει αρχίσει να μελετά την κλιματική αλλαγή. Κυρίως όμως για το δικό του, σε σχέση με το δικό τους ρόλο όσον αφορά την ανταπόκριση στις θεομηνίες για να καλύψουν τα κενά και να προσαρμοστούν. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε είναι κάτι πέραν αυτού. Δηλαδή αφενός χρειαζόμαστε μια ευρύτερη στρατηγική και πολλά που πάθηκαν προηγουμένω είναι αξιόλογα. Δηλαδή να μην ξεκινάμε στις πολιτικές μόνο και να παραμένουμε σε υψηλό επίπεδο αλλά και στο πιο χαμηλό επιτόπου. Θα πρέπει λοιπόν οι στρατιωτικοί να καταλάβουν ότι η κατανόηση της κλιματικής αλλαγής θα βοηθήσει τις ε, πολιτικές ασφάλειας και ε, στρατικές πολιτικές. Δεν είναι κάτι αμεληταίο. Μιλάμε για την σύγκληση τεράστιων τάσεων παγκοσμίω, αύξηση του πληθυσμού, κλιματική αλλαγή, σειράξει. Μιλάμε σφαιρικά για αυτού του κινδύνου και γι' αυτό ακριβώ αυτή η στρατηγική σκέψη είναι απαραίτητη. Αυτό σημαίνει, όσον αφορά το σχεδιασμό, ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον στρατηγικό σχεδιασμό. Θα πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις έχει αυτό πρακτικά, αλλά, να δούμε αν θα πρέπει να έχουμε και ένα σύστημα αγκές το οποίο θα εντάξει και κλιματικούς παράγοντες στα συστήματα αγκές Να καταλήξω λέγοντας ότι θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία των παραγόντων και φορέων ασφαλείας ώστε αυτοί να αποτελέσουν τους πρεσβευτές αυτών των κινδύνων, να μιλήσουν ανοιχτά και να τους λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καθηγητής ε, κύριος Τόρ Μπεν Ιάμινσεν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Okay. <clears throat> Thank you very much. And... Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πραγματικά τιμή μου που έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω για αυτό το σημαντικό θέμα. giving this talk. Ε, ποιο είναι το ιστορικό και το υπόβαθρο από τα τέλη της δεκαετίας του 80 έχω κάνει έρευνα στο Μάλι, στη Δυτική Αφρική, γιατί θα σας μιλήσω για την ασφάλεια του κλίματος στην περιοχή του Σαχέλ. Στην αρχή ασχολήθηκα με την απερίμωση και γενικότερα με τις συγκρούσεις για την ιδιοκτησία της γης. Ξέρετε ότι κυριαρχεί αυτό στην ε, παγκόσμια πολιτική σήμερα και ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η κλιματική αλλαγή. Ακούσαμε σχετικά προηγουμένως. Ε, η περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική ε, συχνά αναφέρεται ως χαρακτηριστική περίπτωση ε, περιοχής που υπάρχουν σειράξεις λόγω κλιματικών δύσκολων. Αναφέρθηκε η λίμνη Τσάντ προηγουμένως. Θα ήθελα να σας δώσω αμέσως το βασικό μου επιχείρημα και τι θέλω να πω. Γενικά εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου για αυτή ε, την συλλογιστική και θα σας εξηγήσω γιατί βεβαίως η κλιματική αλλαγή είναι πολύ επικίνδυνη και θα πρέπει να την πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη. that in... Αλλά ε, έχει δείξει η προϊστορία ότι οι συγκρούσεις και η βία στην περιοχή του Σαχέλ προκαλούνται για άλλους λόγους, πολιτικούς και ιστορικούς. With climate... Και το πρόβλημα που έχουμε εκεί, ε, αν ε, τα φορτώσουμε στην κλιματική αλλαγή, είναι το εξής παραγνωρίζουμε, εξεχνούμε ε, τις πραγματικές αιτίες, όπως είναι ο τζιχαντισμός που βλέπουμε σήμερα στη Δυτική Αφρική. Θεωρητικά η κλιματική αλλαγή μπορεί να διαδραματίσει ε, ρόλο, αλλά η εμπειρική, η πρακτική, τι λέει. Μια άλλη ιστορία που θα σας την πω τώρα εγώ. Okay. So, um, Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή έχει τώρα αναχθεί σε θέμα ασφαλείας. Όταν το 2007 ε, δόθηκε το βραβείο Νόμπελ, αναφέρθηκε η Επιτροπή η Νορβηγική σε αυτό το θέμα, ε, στους κλιματικούς λεγόμενους πολέμους, έχουν ε, εκδοθεί κάποια βιβλία πρόσφατα ε, και ακούμε ότι το κλίμα δεν είναι αυτό καθ' αυτό αιτία πολέμου, αλλά πολλαπλασιαστή των απειλών και των κινδύνων. Τι σημαίνει αυτό όμως και πώς σοβαρά θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη για να θεωρηθεί και πολλαπλασιαστής απειλών. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο πολλές φορές στη συζήτηση. Uh, λοιπόν, αυτό είναι το εξώφυλλο ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε πέρσι. Όταν συζητούμε την ασφάλεια του κλίματος στη Σαχέλ, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι η επίπτωση και ποιος είναι ο αντίκτυπος και συχνά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή οδήγησε ε, στην ξηρασία και στην απερίμωση συμβαίνει πραγματικά περίμωση με αξιόλογο και σημαντικό τρόπο. Αυτό είναι το ερώτημα. Το συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν, το οποίο δημοσιεύθηκε το 2016, αναθεωρεί ε, την διεθνή έρευνα που έχει γίνει για την απερίμωση και ε, περιληπτικά αναφέρει τα σημαντικότερα ευρήματα. Και ουσιαστικά έχει πρασινίσει η ε, περιοχή ε, μετά τις ξηρασίες του 1980. Ενώ λοιπόν συζητούν οι επιστήμονες για πρασίνισμα και πώς συνέβη στην περιοχή του Σαχέλ τις τελευταίες δεκαετίες, τα μίντια και οι πολιτικοί συζητούν ακόμα για απερίμωση και για ξηρασία κλπ. Να σας δώσω κάποιες εικόνες από το Βόρειο Μαλί, κάποιες φωτογραφίες για να καταλάβετε πόσο πρασίνησε ο τόπος. Ε, αυτές οι φωτογραφίες είναι ε, με το ίδιο πλαίσιο, στο ίδιο μέρος και θα σας δείξω την ετήσια εξέλιξη. Ο Θιερή Αγνώ, ένας συνάδελφός μου, ε, ερευνητή στην Τουλούζη, στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών, ΣΕΝΕΡΕΣ, κάνει ε, έρευνα στη Σαχέλ και άρχισε λοιπόν να παρακολουθεί την αλλαγή της βλάστησης στο Βόρειο Μάλι στην αρχή του 80. Εδώ είναι το 1984, βέβαια στην περίοδο των βροχών, Σημειώνω ότι το 84 ήταν η χρονιά με τη χειρότερη ξηρασία από όλη τη δεκαετία του 80 στο Σαχέλ. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που βρέχει περισσότερο εκεί. Πολύ κακή χρονιά. Βλέπετε λοιπόν τον Αύγουστο του 1984 με πάρα πολύ μικρή βλάστηση. Το χόρτο είναι πολύ λίγο. Θα βλέπετε πάντα το ίδιο δέντρο δεξιά. 85 πάλι κακή χρονιά, περίοδος βροχών, λίγο παραπάνω πράσινο ε, και χορτάρι. Το 1988 πάρα πολύ καλή χρονιά. Το 89, όχι τόσο καλή. Το 92, καλούτσικη. Και το 99, εξαιρετική. Βλέπετε λοιπόν πόσο έχει πρασινίσει και η περιοχή και συνεχίζεται αυτό από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Ε, αυτό φαίνεται και από ε, τους δορυφόρους, αν μελετήσετε τις δορυφορικές φωτογραφίες γεωγράφοι ε, στο Πανεπιστήμιο του Λούντ στην ε, Σουηδία έχουν συγκρίνει δορυφορικές φωτογραφίες από το 82 μέχρι το 99. και δείχνει πόσο έχει πρασινίσει το Σαχέλ από τότε, από τις μεγάλες ξηρασίες δεκαετίας του 80. Uh, so, so rainfall has increased. Άρα οι βροχοπτώσεις έχουν αυξηθεί γιατί το πρασίνισμα με αυτό συνδέεται. Πέφτει περισσότερη βροχή και έχει πιο πολύ πράσινο. Ε, αποφάσισα να σας δείξω λοιπόν ε, τις βροχοπτώσεις στο Ντακάρ. Βέβαια το Ντακάρ δεν είναι ακριβώς ε, χαρακτηριστική περιοχή του Σαχέλ, αλλά ίδιες βροχοπτώσεις έχει και ίδιο σχήμα και καιρικέ συνθήκες. Και εδώ βλέπουμε την εξέλιξη. Αποφάσισα να διαλέξω τον Ντακάρ γιατί ε, από τη Δυτική Αφρική ε, καταγράφονται από πολύ παλιά οι βροχοπτώσεις, ετήσιες βροχοπτώσει και ο μέσος όρος πενταετίας από το 1800 παρακαλώ 95 μέχρι το 2015. Και αυτό δείχνει τη γενικότερη τάση που παρατηρούμε και στη συνολική περιοχή του Σαχέλ. Ήταν πολύ καλές οι βροχοπτώσεις ε, στη δεκαετία του 50 κυρίως, 70 και 80 πολύ ξηρή περίοδος, μεγάλη λειψιδρία και σιγά σιγά αυξήθηκε και τουλάχιστον ε, μια μερική ανάκτηση του επίπεδου των βροχοπτώσεων παρατηρήθηκε σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Άρα, παρά το γεγονός ότι είναι πιο πράσινη η περιοχή του Σαχέλ σήμερα από ό,τι ποτέ στο παρελθόν, συχνά ακούμε ε, και διαβάζουμε σε blogs ότι η βία στην περιοχή συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Εδώ έχουμε ένα άρθρο από τη γαλλική εφημερίδα Le Monde και αναφέρεται στην εξέγερση ως ε, ε, ε, το τζιχάτ των φουλάνι που είναι μια εθνοτική ομάδα εκεί και θεωρούν ότι εν μέρει αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Και ξαφνικά λοιπόν στο Μάλι, μάλλον δυστυχώς, θα γνωρίζετε ότι διάφορες τζιχατιστικές ομάδες ελέγχουν το κεντρικό και το βόρειο Μαλί, ενώ οι πόλεις, μόνο οι πόλεις ελέγχονται από το κράτος και το στρατό. Συνεπώς, um, τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι μικροί ε, αγρότες και βοσκοί κυρίως έχουν ενταχθεί σε αυτές τις διχατιστικές ομάδες. Γιατί? Η κλιματική ε, αλλαγή δεν έχει επηρεάσει ε, τις περιουσίες τους. Αλλά πολύ συχνά η, κρατική πολιτική με τη βοήθεια της δύση έχουν περιθωριοποιήσει τον κόσμο. Άρα οι βοσκοί χάνουν την πρόσβαση σε ε, βοσκοτόπια στην ξηρή περίοδο και οι δρόμοι που παίρνουν τα κοπάδια ε, κόβονται λόγω της ε, γεωργικής ανάπτυξης και της γεωργίας. Δηλαδή χάνουν την πρόσβαση στους βοσκοτόπους ε, και τους διαδρόμους που περνούν τα κοπάδια τους ε, λόγω της γεωργικής ανάπτυξης. Γιατί δίνουν εκεί την έμφαση και ευνοούν τη γεωργία ε, και εις βάρος της κτηνοτροφίας που είναι εκτατική σε βοσκοτόπους και πλανόδια. Αυτό ισχύει για το Μάλι αλλά και για το Σαχέλ. Δεύτερον, η διαφθορά ε, αυξήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ε, και στη διοίκηση και στη δικαιοσύνη. Ε, και αυτό ενέτεινε το θυμό μεταξύ των γεωργών και των αγροτών, γιατί υπάρχουν μεγάλες συγκρούσεις ως προς την ιδιοκτησία της γης και γι' αυτό, αυτό όξινε και τα αισθήματα του κόσμου κατά του κράτους, κατά των ελίτ, κατά της κυβέρνησης. Και είναι πολύ πονηροί οι και τα εκμεταλλεύονται αυτά τα ε, αισθήματα του κόσμου και τις ε, δυσφορίες. Αυτά η διεθνή κοινότητα δεν τα καταλαβαίνει. Έχει τελείως παραγνωρίσει αυτό το γεγονός. Ενώ το Μάλι ε, ήταν ένα υπόδειγμα δημοκρατικής ανάπτυξης. Μέχρι να αρχίσει η κρίση το 2012 το παρουσίαζαν διεθνώς ως ένα υπόδειγμα για την Αφρικανική Δημοκρατία. Πολύ ενδιαφέρον αλλά και πολύ περίεργο ταυτόχρονα να διαπιστώνει κανείς ε, αυτή την αντίθεση, αυτή τη σύγκρουση για το πώς ε, παρουσίαζαν το Μάλι διεθνώς, ε, ενώ το, αυτό που συνέβαινε στη χώρα ήταν συζητήσεις για την κρίση της δημοκρατίας στη χώρα και για την αύξηση της διαφθοράς. Άρα, για ποιο λόγο λοιπόν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ε, πήγαν σε τις τζιχαθιστικές ομάδες. Μελέτησα ε, τις ομιλίες του Χαμαντών Κούφα, ο οποίος θεωρείται γενικά ο ύψιστος ηγέτης των τζιχαντιστών στο κεντρικό Μάλι. Και τι λέει λοιπόν στις ομιλίες του. Κατηγορεί κυβερνητικούς ε, υπαλλήλους, δικαστικούς και την ελίτ και την κρατική αλλά και τον φυλάρχων για ε, ευρεία διαφθορά και ε, κακοδιαχείριση και είναι υπέρ ε, της ισότητας και της εκτατικής γεωργίας και εκτινοτροφίας και των βοσκών ως τρόπο ζωής και διαβίωσης. Έτσι λοιπόν, τι είναι αυτό που προκαλεί συγκρούσεις για τη χρήση γης στο Σαχέλ. Εκ των ιδίων μου ερευνών έχω καταλήξει, βέβαια και συνεργασία με συναδέλφους, σε κάποια συμπεράσματα, ε, τα οποία θα ήθελα να σας αναφέρω. Πρώτον, υπάρχουν πολιτικές και νομοθεσία που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. αποκλείονται οι βοσκοί από κάποιους διαδρόμους, από κάποια χυμαδιά ας πούμε που πηγαίνουν και βόσκουν τα ζώα τους στην ε, περιοχή της ξηρασίας. Και επίσης υπάρχει και η διαφθορά η οποία υπονομεύει ε, την εμπιστοσύνη και ε, την πίστη του κόσμου στους κρατικούς θεσμούς. Η κρηματική αλλαγή βεβαίως μπορεί να παίξει ρόλο, αλλά μέχρι τώρα είναι δύσκολο να εντοπίσουμε σαφή αντίκτυπο ε, ξέρουμε ότι αυξάνονται οι θερμοκρασίες, ωραία. Αλλά δεν γνωρίζουμε ε, πώς ε, οι βροχοπτώσεις ε, και η περιοδικότητά τους επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν κλιματικά μοντέλα σήμερα τα οποία προβλέπουν περισσότερες βροχοπτώσεις, όχι λιγότερες και πιο συγκεντρωμένες. Άρα αλλαγές θα υπάρξουν στο κλίμα, στο σαχέλα. Αυτό πώς θα επηρεάσει τη χρήση γης δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ε, θα επηρεαστεί η κατάσταση από την κλιματική αλλαγή και μπορεί να ενταθούν οι συγκρούσεις εκεί και οι εντάσεις ακόμα περισσότερο. Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι μέχρι τώρα οι πολιτικές αιτίες είναι πολύ πιο εύγλωτες για να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις και οι ταραχές στο Μάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μάλιν Μπόμπιορκ. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Thank you so much. Από το Σύπρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Πραγματικά μετά από μία ώρα ε, είναι μεγάλη πρόκληση να πω και εγώ κάτι ε, διαφορετικό. Χαίρομαι πολύ πάντως που είμαι εδώ. Εγώ δουλεύω στο ΣΥΠΡΙ που είναι το Διεθνές ε, Ειρηνευτικό Ίδρυμα της Στοχόλμης και θα ήθελα να αναφερθώ στη δουλειά μας που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα ήθελα να δώσω και μια ευρύτερη ε, θεώρηση άλλων ε, θεμάτων που καλύπτουμε στο ΣΥΠΡΙ ε, έχει να κάνει με θέματα όσον αφορά την ενίσχυση και την αύξηση της, γνώμης μας, της γνώσης μας μεταξύ της ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής. Είναι ένα περίπλοκος τομέας που εξελίσσεται πολύ και η δική μας προσπάθεια ήταν ουσιαστικά προσπαθήσαμε να δούμε τις διόδους ε, μεταξύ της ασφάλειας και των ε, βίαιων συγκρούσεων και της κλιματικής αλλαγής. Οι βίαιες συγκρούσεις έχουν πάντοτε ε, κάποια πολιτική και ιστορική διάσταση, όμως πώς και υπό ποιες συνθήκες οι αλλαγές που προέρχονται από το κλίμα και το ίδιο το κλίμα μπορεί να επηρεάσουν αυτές τις συνθήκες. Είναι κάτι που θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Ένας ακόμη τομέας επί του οποίου εργαζόμαστε είναι διεθνείς ε, οργανισμοί και πώς ε, αντιδρούν σε ε, κινδύνους ασφαλείας προερχόμενους από το κλίμα. Οργανισμοί όπως ο ΙΕ, η ΑΣΕΑΝ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί Υπάρχουν βέβαια και αναλύσεις ε, ειδικέ αναχώρα, ε, οι οποίες και αυτές ε, παίζουν το ρόλο, γιατί Προφανώς υπάρχουν ε, και κάποια εθνικά συμφέροντα που επηρεάζουν ε, ευρύτερα τους οργανισμούς οποίους ανήκουν, αλλά και οι οργανισμοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ε, στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση όλων αυτών των κινδύνων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, θέλουμε να συνεισφέρουμε ε, στην ανάπτυξη, στην ύπαρξη βοήθειας, να μπορέσουμε να ανταποκρινόμαστε γρηγορότερα ε, στις ανάγκες και να μπορέσουμε να ε, παρέχουμε καλύτερες συστάσεις για το πώς μπορούμε να μετριάσουμε τους κινδύνους και να τους προλάβουμε. Όσον αφορά την πολιτική, ε, έχουμε πολλούς εταίρους όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικής ε, και, ε, και με ακαδημαϊκούς και επιστήμονες. Με τον Νίκολας Μπρίμς συνεργάζομαι πάρα πολύ από το Σουηδικό Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων. Μπορείτε να έρθετε και σε επαφή μαζί του αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, έχω και μερικές διαφάνειες. Λίγο περισσότερα θα ήθελα να πω σε σχέση με τις προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας ε, και τη σχετική πολιτική. Κάποιοι από τους συναδέλφους ήδη ανέφεραν ορισμένα πράγματα γι' αυτό. Θα ήθελα όμως και εγώ να πω, ε, να κάνω κάποια σχόλια. Ε, γνωρίζουμε πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την κατάσταση. Η δυναμική των συγκρούσεων είναι σημαντική. Υπάρχει μια διάκριση που πρέπει να γίνει ε, ανάμεσα στους, στις αιτίε και στη δυναμική ε, η οι λόγοι μπορεί να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να την προλάβουμε, όμως η κλιματική αλλαγή έχει να κάνει και με τη δυναμική ε, συγκρούσεων οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει και πώς μπορούμε να τις σταματήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στην κατανόηση, του, είναι λοιπόν πολύ σημαντική η κατανόηση του πώς το κλίμα επηρεάζει αυτές τις συγκρούσεις. Δεν επηρεάζει όλες τις ε, ε, συγκρούσεις. Ε, προφανώς στην υποσαχάρια Αφρική τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Καταλαβαίνω περισσότερα, καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετική η κατάσταση στην Ανατολική Αφρική για παράδειγμα. Πάντως σε μερικές περιοχές η σύνδεση μεταξύ των δύο είναι πολύ έντονη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό από άποψη ασφάλεια αλλά και στις σε τι διεθνεί σχέσει πώ εκφράζεται αυτή η σχέση μεταξύ κλιματική αλλαγή και ασφάλεια και άμυνα. Ε, σε τουλάχιστον 120 χώρες έχει γίνει η αναγνώριση του κατά πόσο η κλιματική αλλαγή ε, είναι ένα σημαντικό τμήμα της δικής τους πολιτικής στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η ασφάλεια έχει να κάνει όμως και με τη θε, ε, θεώρηση των πραγμάτων. Έχει σημασία δηλαδή το πώς βλέπουμε το μέλλον και έχει σημασία πώς επηρεάζονται και οι σχέσεις, η, τα τρόφιμα, η ενέργεια, το νερό. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Τρίτο τομέας, πώς επηρεάζει δηλαδή τις διεθνείς αποστολές ε, όσον αφορά του τι είδους αποστολή είναι είναι ε, τι περιβαλλοντικές ε, ε, αποστολές λαμβάνουν χώρα στην περιοχή και τι κίνδυνοι υπάρχουν ασφάλειας και άμυνα στη συγκεκριμένη περιοχή αυτή. τρεις λοιπόν τομείς είναι τομείς στους οποίους παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το κλίμα και συνδέεται με την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Με αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αλλάξει και η πολιτική που θα ακολουθηθεί. Έχουμε δει την αξιολόγηση κινδύνων, την πρόληψη, όλη αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση, όλες αυτές ε, οι εμβληματικές λέξεις στις οποίες αναφερόμαστε συνεχώς. Θα το εξηγήσω και αυτό σε λίγο. Λοιπόν, να επικεντρωθώ περισσότερο στην ε, ε, πολιτική κλίματος και ασφάλειας και το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάμε λίγο προς τα πίσω για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Να αρχίσουμε λοιπόν με το να δούμε ε, ποια είναι η ιστορία ε, του πράγματος. Ε, είναι κάτι το οποίο ίσως αναφέρθηκε ήδη, αλλά η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Το 2008 το έγγραφο Σολάνα για την κλιματική αλλαγή και την εθνική ασφάλεια είναι ένα ε, βασικό έγγραφο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αρχίσει ε, η δουλειά στον τομέα αυτό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έγγραφο αυτό υπήρχε αυτή η έννοια του πολλαπλασιαστή απειλής, εμφανίστηκε για πρώτη φορά την ίδια χρονιά, το 2008, έγινε μια ενημέρωση της προηγούμενης ε, στρατηγικής ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία άλλαξε τον τόνο και αναγνώρισε σαφώς ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλώς μια παγκόσμια ε, πρόκληση, είναι μια βασική απειλή στα ευρωπαϊκά συμφέροντα και αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό ε, και και στις απειλές εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, ε, αλλά επηρεάζει τα συμφέροντα ασφαλείας ε, της Ευρώπης. Μετά, ε, ένα μεγάλο μέρος της εργασίας ξεκίνησε τότε Όμω, επειδή απέτυχαν οι συνομιλίε στην Κοπενχάγη για το περιβάλλον, κάπως ε, έπεσε το επίπεδο των φιλοδοξιών και το ηθικό ε, σε διάφορες χώρε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όμως συνέχισαν, συνέχισε να γίνεται κάποια δουλειά που αποτελεί το θεμέλιο της δουλειάς που γίνεται σήμερα. Για παράδειγμα, Λισαβόνα το 2009, γιατί άρχισε να, βλέ, να, να, να είναι διαφορετική η θεώρηση της πολιτικής ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ ευρύτερο τρόπο ότι πηγαίνει πέρα από την ε, ε, συνεργασία ε, ε, στρατιωτικού πολιτικού τομέα και αυτό άρχισε να τίθεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και τι γίνεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπήρχε ε, η ατζέντα του 2030 και η Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή που επίσης δημιουργεί ένα πλώσιο για το πώς ε, πρέπει να προχωρήσουμε, οι στόχοι της αηφόρου ανάπτυξης, πώς μπορούμε δηλαδή να συνδυάσουμε πολλούς τομείς Κάτι το οποίο φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά, πέρσι ήρθε ε, η στρατηγική ασφάλεια Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πέρσι Βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι τμήμα της κατανόησης της στρατηγικής, μεταξύ άλλων πτυχών βέβαια που είναι πολύ σημαντικές, ε, ε, με την ευρεία έννοια της, της ασφάλειας πλέον για την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, Τι τονίζει αυτή η στρατηγική ασφαλείας, για παράδειγμα, πώς η κλιματική αλλαγή είναι μια πτυχή που μπορεί να διακυβεύσει ε, την κατάσταση, να είναι επικίνδυνη για τους πολίτες και για το έδαφος, ότι επίση η αλλίωση του εδάφους και του περιβάλλοντος μπορεί να επιδεινώνει ενδεχόμενες συγκρούσεις ε, λόγω του αντικτύπου, στην απερίμωση, ε, την διάβρωση του εδάφους, την, την λειψιδρία και την έλλειψη τροφίμων Όλα, ε, επίσης ε, και ε, είναι πάρα πολύ σημαντική και η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και να τα αμβλύνει είναι η πρόληψη. Η πρόληψη είναι πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να επικεντρωθούμε στις βασικές αιτίες, γίνεται πολλή δουλειά σχετικά και στο, στον ΟΗΕ, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίες. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει μια λοιπόν πολύ ευρία θεώρηση του τι είναι ασφάλεια, ε, ότι υπάρχουν πολλές πτυχές που την επηρεάζουν και επίσης προκειμένου να μετριάσουμε όλους αυτούς τους επιβαρυντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια, ένα από αυτά ε, είναι τα τρόφιμα. Είναι φυσικά και μια τεράστια πρόκληση. Πώς είναι δυνατόν να ε, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της έλλειψης τροφίμων. Κάτι το οποίο ε, ολοκληρώθηκε πέρσι, ε, μία μελέτη περιπτώσεων ή τέλο πάντων εστιασμένη ανάλυση για το πώς η ΕΙΕΔ ε, άρχισε να λαμβάνει υπόψη της τα θέματα του κλίματος. Υπήρχε μάλιστα και ένα συγκεκριμένο πόρισμα εγώ είχα κάποιε επιφυλάξει να σα πω την αλήθεια, γιατί από τότε που υπήρξε αυτή η στρατηγική της ε, ασφαλείας έχει γίνει πολλή δουλειά στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω κάποια παραδείγματα και θα σα πω ε, κάποιους από του προβληματισμού μου που πιστεύουμε ότι οδεύει όλο αυτό. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη λοιπόν μεμονωμένη περίπτωση που εξετάστηκε η, εστιασμένη ε, ε, αυτή η ανάλυση για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι νομίζω ενδεχομένω ε, σημαντικό να το σκεφτούμε. Λοιπόν, Είχαμε συνεντεύξεις, επαφές ε, με σημαντικούς αξιωματούχους και ανθρώπους που δουλεύουν πολύ κοντά στην ΕΙΕΒ. Όσον αφορά τις προκλήσεις, όταν ε, ιδρύθηκε η ΕΙΕΒ, άρχισαν να, να δημιουργούνται και νέες μορφές συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α, ε, τομείς που δεν είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν άρχισαν να συνεργάζονται και αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο γιατί υπάρχουν διαφορετικές εντολές, διαφορετικές παραδόσεις, ε, ε, ε, τρόποι αντίληψης των πραγμάτων. Η ΕΕ λοιπόν διαδραματίζει ένα ρόλο και προσπαθώ, προσπαθεί να ε, συντονίσει τις μεμονωμένες εργασίες των διαφόρων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η γεφύρωση, εν πάση περιπτώσει, των διαφορών και ο συντονισμός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει κάποια πρόχειρη λύση που να μπορούμε να βρούμε. Ε, υπάρχει μια προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί. Υπάρχει λοιπόν μια ανισορροπία μεταξύ της ικανότητας ε, αντιμετώπισης αυτών και επεξεργασία αυτών των θεματικών ε, ενωτήτων που μερικές φορές είναι μακροχρόνια ζητήματα. Αποκινούμε άλλους φορείς ε, που είναι πολύ ευρύτεροι γιατί υπάρχουν αρκετοί εμπειρογνώμονε για την ε, ε, κλιματική ε, ασφάλεια. Πρέπει δηλαδή κάποιο να είναι εμπειρογνώμων για να μπορεί να καταλάβει περί τίνο ακριβώ πρόκειται. Υπάρχει λοιπόν μια ανισορροπία μεταξύ των διαφόρων φορέων ω προ την ικανότητά του να συνεργαστούν. Όσον αφορά τώρα την περιεκτική και συνολική προσέγγιση, ναι, πράγματι είναι πολύ σωστή η κατανόηση πλέον σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω Υπάρχει μια εστίωση στην αντίδραση, στην αντιμετώπιση των κρίσεων σε βραχυπρόθεσμες προσεγγίσεις ε, εφαρμογής. Η, η πλευρά της αντίδρασης είναι ισχυρότερη δηλαδή, παρά το γεγονός ε, ότι η πρόληψη αναφέρεται στα χαρτιά. Στην πράξη όμως δεν γίνεται αυτό. Ένας τρίτος τομέας ε, είναι ότι η ασφάλεια δεν είναι μια απλή έννοια είναι δύσκολο να υπάρχει μια ενιαία θεώρηση του τι θα πει ασφάλεια. Μερικές φορές θεωρεί κανείς ότι η ασφάλεια είναι κάτι, μια στρατιωτική έννοια. Δεν σημαίνει ότι ο στρατιωτικός τομέα έχει το βασικό ρόλο να ε, ε, ε, εξασφαλίζει την ασφάλεια. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος ε, να ε, συζητήσουμε με διάφορου φορεί που έχουν μια διαφορετική θεώρηση τη ασφάλεια και αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνει. Όσον αφορά τώρα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αυτή η κλιματική διπλωματία, αυτό το δίκτυο κλιματικής διπλωματίας για την πράσινη δημοκρατία, το, ε, συγγνώμη, διπλωματία για την πράσινη διπλωματία, το δίκτυο πράσινης διπλωματίας, είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι υπαρκτό, θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα ρόλο, αλλά δεν το κάνει στην πραγματικότητα. Και εδώ νομίζουμε Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το δίκτυο πρέπει να, να διδραματίσει έναν καλύτερο ρόλο. Όσον αφορά τώρα την ανθεκτικότητα των αποστολών ε, των ειρηνευτικών. Είναι κάτι δύσκολο βέβαια γιατί η πρόληψη των κρίσεων σε έναν οργανισμό που περισσότερο επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ε, ήδη μενωμένων ε, συγκρούσεων είναι δύσκολο υπάρχει και ο τομέας αναπτυξιακής πολιτικής και ίσως μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας να μπορεί κανείς να αναπτύξει αυτή την ανθεκτικότητα που λείπει. Ένας, μία από τις σκέψεις μου για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση είναι η, πραγματικά το να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανθεκτικότητα. Πώς μπορούμε δηλαδή να την, να την κάνουμε πραγματικότητα. Οι περισσότεροι ενδεχομένω στην αίθουσα αυτή γνωρίζουν περισσότερα για το τι ακριβώ γίνεται από απόψε ω ε, σχεδίων και προγραμμάτων ε, ω προ τον τομέα αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο. Ε, ε, της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά χρειάζεται μία αξιολόγηση κινδύνου ε, σε σχέση με το κλίμα. Ε, προφανώς γίνεται αυτό, έχει δρομολογηθεί, αλλά χρειάζεται να γίνεται πολύ πιο συστηματικά και υπάρχει επίσης η ανάγκη ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Γιατί η κίνδυνοι του κλίματος είναι τόσο πολύ. Υπάρχει ένα συστημικός κίνδυνο. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν ε, ε, θεματικές ενότητες κινδύνων και να, ε, να κάνετε μια ιεράρχηση από πού πρέπει να ξεκινήσετε και πού πρέπει να φτάσετε ότι είναι ενδεχομένω λιγότερο περίπλοκο να καλυφθεί πιο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει κανείς να αναπτύξει μία υποδομή, πρέπει να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές του. Επίσης, υπάρχει η έγκαιρη προειδοποίηση και αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ε, ε, εστίαση στην ε, ικανότητα έγκαιρης προειδοποίησης. Αλλά αν κατάλαβα καλά, από απόψεως κλιματικής είναι πολύ βραχυπρόθεσμη. Νομίζω ότι είναι δύο μήνες περίπου. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συνδέσουμε με την προληπτική δράση που παίρνει ένα χρόνο και μετά μπορείτε να πάτε και πιο πίσω, δηλαδή να αρχίσετε μερικά χρόνια πριν την πρόληψη. Πρέπει λοιπόν να συζητηθεί αυτό σε επίπεδο στρατηγικό με την ηγεσία. Αυτή η στρατηγική ηγεσία, το βλέπουμε αυτό από την εμπειρία μας σε άλλους ε, διεθνείς οργανισμούς, είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Είδα ότι πολλούς από τους τομείς ε, και το λέω αυτό σε σχέση με την εφαρμογή μετά τα πρώτα χρόνια της ε, στρατηγικής ε, της ε, ασφάνειας. Ο άξονας εσωτερικός-εξωτερικός. Αν σκεφτεί κανείς τη σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού, θα μπορούσε αυτό να συμπεριλαμβάνει τη διάσταση, την κλιματική, έχει να κάνει με τη μετανάστευση, έχει να κάνει με το περιβάλλον. Να προσπαθήσει δηλαδή να δεις σε ποιου τομεί μπορεί να αυξήσει τη βαρύτητα του κλίματο. Πρέπει εσεί να δείτε πώ είναι δυνατόν αυτά να τα συμπεριλάβετε στη δουλειά σα. Νομίζω ότι υπάρχει το πλαίσιο το έχετε δημιουργήσει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να καταστεί λειτουργικό εντό του συστήματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα αρχίσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Βαλέρο, η συντονιστριά μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά. Θα πρέπει να βάλετε τα ακουστικά, λοιπόν. Αρχικά να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες που πήραν το λόγο γιατί αυτά που είπατε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ελπίζω η γραμματεία να μας δώσει και τις φωτογραφίες σας γιατί είναι σημαντικό να έχουμε έτσι και μια ανάμνηση φωτογραφική δικιά σας. Τα είχαμε λοιπόν προηγουμένως ότι αυτή η κλιματική αλλαγή έχει διάφορες επιρροές στην ασφάλεια ανάλογα με την περιοχή. Στην Αφρική, ας πούμε, στις στοχές ε, χώρες έχει συγκεκριμένη επιρροή, διαφορετική στην Ακτική. Επίσης, στην Συρία θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα τμήμα της σύραξης οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Στη Σομαλία, ας πούμε, επίσης. Εγώ πήγα στο Μάλι όταν θεωρούταν υπόδειγμα δημοκρατίας. Πήγα εκεί λοιπόν για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να χτίσουμε ένα δημοκρατικό κράτος στην Αφρική. Και ταυτόχρονα ήταν μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου το Μάλι. Αλλά είχαμε αυτές τις υποβόσκουσες σειράξεις μεταξύ του ΑΡΕΚ και του υπόλοιπου πληθυσμού. Αυτές οι ράξεις ήταν πάντοτε παρούσες στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν επίσης και οι διαδρομές που ακολουθούν οι έμποροι ναρκωτικών από την Λατινική Αμερική μέχρι τη Δυτική Αφρική. Υπάρχουν λοιπόν πολλά στοιχεία εδώ για τα οποία δεν πολύ συζητάμε ή δεν πολύ συζητούσαμε επειδή απλά και μόνο θέλαμε να τονίσουμε το θέμα της ε, ειρήνης ή της παρουσίας ειρήνης στο Μαλί. Οπότε αφήναμε τα άλλα κατά μέρος. Για αυτά που είπατε για την μετεωρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλοί οικολόγοι που βρίσκονται στη χώρα αυτή στο Μάλι και είμαι σε τακτική επαφή μαζί τους και μέσω ενός σωτικού προγράμματος βοήθειας μπόρεσα να πάω εκεί, σε αυτή τη χώρα και είδα πραγματικά ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που συνδέονται με την κλιματική αλήγη και υπάρχει μια ουσιαστική δουλειά που γίνεται ώστε να μην διαδοθεί αυτή η κρίση. Γίνεται λοιπόν μια δουλειά για να αποτραπεί η απερίμωση και μάλιστα πήγα σε ένα μικρό χωριό, μίλησα με τους κατοίκους που μας είπαν ότι ανέκαθεν ήταν γεωργοί και κοίταζαν τον ουρανό. Όταν έβλεπαν λοιπόν τα αποδημητικά πουλιά να έρχονται, τότε αμέσως ψαχνάν ε, προστασία γιατί ήξεραν ότι έβρεχε αμέσως. Τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Ή δεν έρχεται καθόλου η βροχή ή έρχεται ταυτόχρονα με τα αποδημητικα Η βροχή λοιπόν πάντα υπάρχει, υπάρχουν βροχοπτώσεις, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε όπως παλαιότερα πότε θα συμβούν. Αυτό έχει επιπτώσεις στην καλλιέργειες, στη φτώχεια και στην κατάσταση δηλαδή στην εσωτερική αυτής της χώρας, στο Μάλι. Και υπάρχουν επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συγκεκριμένε εδώ. Τώρα για το θέμα της ασφάλειας. Πάντοτε στο Μάλι. Στο τέλος της εισηγησής σας είπατε ότι δεν μπορούμε πάντοτε με στρατιωτικό τρόπο να λύνουμε τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Μπορεί ίσως και κάποιες χώρες φτωχές, αλλά για μας κάποιες απειλές που αφορούν ας πούμε υποδομές ή και πολλά άλλα πράγματα που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή δεν, δεν μπορούμε να τα θα αντιμετωπίσουμε άμεσα όλα αυτά. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε τι ε, κοινωνίε μα για τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή, Εδώ και χρόνια το κάνουμε αυτό στη Σουηδία. Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια τεράστια απειλή για την ασφάλεια της ίδιας της χώρας, της Σουηδίας. Και τώρα πια μιλάμε για την ασφάλεια των ατόμων και την ασφάλεια της χώρας. Ξεκάθαρα. Θα ήθελα λοιπόν και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτά τα θέματα. Δηλαδή, όταν έχουμε να κάνουμε θέματα ασφάλειας, μιλάμε για την ασφάλεια της, των χωρών μας. Αλλά να μην έχουμε ψευδεστήσεις για την ασφάλεια των ατόμων πρόκειται. Αυτό μας αφορά πιο άμεσα. Οπότε θα έπρεπε να έχουμε ένα νέο τρόπο προσέγγισης, ένα νέο τρόπο σκέψης, μια νέα νοοτροπία. Μιλήσατε προηγουμένως για αυτή την αποσπασματική προσέγγιση και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση. Θα πρέπει δηλαδή να αποφύγουμε την αποσπασματικότητα. Όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, μιλάμε εδώ ας πούμε, αλλά σε μια άλλη επιτροπή που ασχολείται ας πούμε με την άμυνα ή με την εξωτερική πολιτική, δεν μιλάνε, δεν μιλάνε για την κλιματική αλλαγή, αλλά μιλούν ενδεχομένω για το περιβάλλον, α πούμε, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά όχι διασυνδέοντάτος απαραίτητα με θέματα ασφάλειας και άμυνας. Θεωρώ ξεκάθαρα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ ασφάλειας και κλιματικής αλλαγής. Ε, θα μπορούσα να σας κάνω και πολλές ερωτήσεις, είχα αυτά τα σχόλια κυρίως, αλλά θα ήθελα να μας στείλετε τις ε, εισηγήσεις να τις έχουμε γραπτώσει. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα μιλήσω αγγλικά παρόλο που είμαι Γερμανός. Και γερμανικά μπορείτε να μιλήσετε. Το πρωί μιλούσατε σε μένα ε, και μου μιλήσατε αγγλικά, αλλά κανονικά όπως θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλώς είναι σας, θα συνεχίσω στα αγγλικά. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων ε, για το πάνελ αυτό που συγκεντρώσαμε σήμερα. Είναι από τα θέματα ε, τα οποία με ενδιαφέρουν και μένα. Ε, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται. Εγώ είμαι Γερμανός σοσιαλδημοκράτης, ανήκω στην ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών και στην ακρόαση της ρώτησα την κυρία Μογκερίνη ποια είναι η αποψή της για την κλιματική διπλωματία απάντησε, εστίασε σε αυτό ότι είναι υπέρ και αναπτύσσει ε, τη διπλωματία και ζήτησε να, υπάρξει και μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για την κλιματική διπλωματία πριν από 1,5 χρόνο. Τώρα ακόμα είναι σε διαδικασία εκπόνησης η έκθεση, αλλά πηγαίνει καλά. Και προσβλέπω να συνεργαστούμε. Πολύ χρήσιμη η ακρόαση και σημείωσα πάρα πολλά. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Έχω πάει δύο φορές ε, ε, στη Νέα Υόρκη. Είμαι μέλος της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Χθες είχαμε μια κρόση με 24 χώρες Αφρικής και ε, το Κοινοβούλιο πραγματικά επενέθηκε για τους στόχους της, ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε. Στις διαπραγματεύσεις εμπορικές με τον Καναδά έχουμε πει ότι θέλουμε να υλοποιηθεί η Συμφωνία των Παρισίων. Είναι ένα νέο μέσο. Εσείς το έχετε κοιτάξει, είναι ενδιαφέρον στοιχείο για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική να το βάζουμε και στις συμφωνίες τις εμπορικές. Χρειάζεται το δίκτυο ε, να στηθεί, να αρχίσει να λειτουργεί, να έχει και ένα μυϊκό σύστημα. Ε, τι γίνεται στην υπηρεσία εξωτερική δράση, υπάρχει κανένα τέτοιο μυϊκό σύστημα να το ενισχύσουμε. Δεν λέω bodybuilding, ας πούμε, να τους κάνουμε και πρωταθλήτε Και ποια είναι η σχέση σας και η συνεργασία σας με την Ηνωμένα Έθνη. Επισκέφτηκα και εκεί και για το κλιματικό πρόγραμμα τους απασχολεί και το αποτύπωμα που αφήνουν τα διάφορα προγράμματα του ΟΗΕ, το ίχνος αυτό το κλιματικό. Και μια τελευταία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εργάζεται με πολλούς συναδέλφους της Επιτροπής ΑΦΕΤ και με Γερμανούς και με Δανό συνάδελφο και μεγάλο για τις κλιματικές αλλαγές και τα θέματα της Συμφωνίας των Παρισιών. Το Brexit είναι επίσης ζήτημα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν πολύ ισχυρή η Βρετανική ε, εξωτερική πολιτική και η κλιματική διπλωματία. Θα τη χάσουμε αυτή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω ε, μπορούμε να προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία γενικές ερωτήσεις. Μπορούμε να διευρύνουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, να έχουμε με ειδικού για το κλίμα. Γιατί το βλέπω και από διάφορες αποστολές που κάνω. Και συνεργαζόμαστε ε, με πόλεις και στην COP23 για πρώτη φορά ήρθε εκπρόσωποι το ΝΟΤΑ. Ε, και της τοπικής και της περιφερειακής αυτοδίκησης Δήμαρχη. μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να εμπλουτίζουμε τις σχέσεις μας με τις πόλεις. Όχι μόνο με κυβερνήσεις. Ζητώ συγγνώμη για τον παράζη των ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις και να πω και κάποια σχόλια. Με την ιδιότητα όμω του κοινού μέλου, όχι τη Πρόεδρου. Μέλο τη Υποεπιτροπή. Ε, θα ήθελα λίγο να σχολιάσω την παρατήρηση της κυρίας Βαλέρο ότι σε διάφορες περιφέρειες του κόσμου η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει διαφορετικές επιπτώσεις ε, στην ασφάλεια πάντα. Εγώ θα πρότεινα να προσθέσουμε κάτι ακόμα ακόμα και στην ίδια περιφέρεια μπορεί να έχει και θετικό και αρνητικό αντίκτυπο η κλιματική αλλαγή. Πάντα για την ασφάλεια. Αρχίζει να μένεις από την Αρκτική. Λιώνουν οι πάγοι, όν οι πάγοι εκεί και αυτό σίγουρα ε, βελτιώνει τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης για μέρη όπως είναι η Γρυλανδία, Φερρυπίν. Έτσι ώστε οι αυτόχθονες ε, πληθυσμοί να μπορέσουν ενδεχομένως να υποφεληθούν από αυτή την αλλαγή. Και με ακαδημαϊκούς όρους μπορεί να είναι ενδεχομένω πολύ θετικό το γεγονός ότι άλλαξε και μια, ε, άνοιξε μάλλον η βόρεια οδός για το εμπόριο μέσω του Βορειού Πόλου. Αλλά βεβαίως υπάρχει πάντα, ιδιαίτερα τέτοιους καιρούς που έχουμε παγκόσμια ε, πολιτική και μετάβαση και μετάβαση ασφαλείας, κάποια ζητήματα. Θυμίζω τις στρατηγικές αναλύσεις ε, του ΝΑΤΟ που θεωρούν ότι οι πρωταγωνιστές εκεί μπορεί να αξιοποιήσουν την κατάσταση και δεν θέλω καθόλου να υποτιμήσω ε, τις αρνητικές συνέπειες για την αύξηση της στάθμης των θαλασσών ε, σε μέρη όπως είναι ο κόλπος της Βενγάλης. Καθόλου παραμένει αυτός ο κίνδυνος. Απλώς ε, δανείστηκα το παράδειγμα αυτό της Αρκτικής για να προσπαθήσω να παρουσιάσω και να φωτίσω και μια άλλη πτυχή. Δηλαδή, η πολιτική συμπεριφορά των πρωταγωνιστών είναι και αυτό ένα ζήτημα. Όχι απλώς κακή, λάθος χρήση γεών εξόριση, αλλά ακόμα και στρατιωτικοποίηση, ας πούμε, αυτών των περιοχών. Και ιστορικά δεν είναι καινούριο. Οι διαστάσεις που έχει προσλάβει μπορεί να είναι, αλλά τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα και αυτές τις απόπειρες και είχαμε και μεγάλους πολέμους. Και γνωρίζουμε ότι είχαν γίνει απόπειρες και στο παρελθόν. When when I look, I must admit... Οφείλω να ομολογήσω, καθηγητά Μίνσεν ότι διαβάζοντας τα βιογραφικά των μελών του πάνελ. Εγώ ήθελα πραγματικά να έχω ε, κάποιον από την Νορβηγία όσο γίνεται πιο επιστημονική προσέγγιση γιατί εδώ και καιρό έχω διαπιστώσει πόσες προσπάθειες κάνουν οι Νορβηγοί, τώρα βλέπω και οι Σουηδοί, οι Σκανδιναβοί γενικώ, να ασχοληθούμε με την αποψήλωση ε, των ε, δασών συγκεκριμένων περιφερειών. Και μάλιστα την αντιμετώπιση της αποψήλωσης, της αναδάσωσης. Βεβαίως χρειάζεται και βοήθεια από τον καιρό. Χρειάζεται βροχή. Αν δεν έχει βροχοπτώσεις δεν γίνεται. Take water for, for, for the whole existence. Οπότε, τώρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο κύκλο και στο Σαχέλ βλέπουμε και κάποια κίνηση ε, στο βόρειο Σαχέλ, ε, στο βόρειο Μάλι. Ε, βλέπουμε κάποιες εξεγέρσεις ακριβώς και λόγω της μετακίνησης και μετανάστευσης των Τουαρέγ από τη Λιβύη, ας πούμε, μετακινήθηκαν προς το Μάλι εκεί υπήρχε και κάποιο εμπόριο όπλων, που μάλλον γι' αυτό το λόγο έγιναν αυτές οι ε, μεταβολές και κόπηκαν κάποιες δίωδοι και για λόγους εσωτερικής πολιτικής αλλά και εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και διάφορα στοιχεία που ποικίλουν. Είναι πάρα πολύ ε, περίπλοκος λοιπόν ο ρόλος αυτών. Δομές βέβαια υπάρχουν, αλλά πώς θα αξιοποιηθούν, αυτό είναι το ζητούμενο. Και είναι σημαντικό να συνδεθεί άμεσα με την ε, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Υπάρχουν πολύ έντονες ε, σειράξεις, πολύ βίες με μεγάλες μετακινήσεις. Όπως είναι στην Ανατολική Ουκρανία υπάρχει τεράστιος κίνδυνος οικολογικής ε, ρήπανσης και ενδεχομένων κλιματικών αλλαγών. Και αλλού. Uh, in terms to, Και θα πρέπει να προλαμβάνονται τέτοιου είδους σειράξεις έτσι κι αλλιώς, αλλά και η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, για παράδειγμα. When we speak about Syria, it's not only it's chemical weapons as well. Δεν είναι μόνο η ξηρασία, που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος και χημικά όπλα. Λοιπόν, υπάρχουν και πολιτικές που ακολουθούν οι διάφορες χώρες, εξωτερική και εσωτερική. Θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα θέματα, αλλά πάρα πολύ δύσκολα να διαρθρωθούν. Και ίσως με την ίδια σειρά. Παρακαλώ, κύριε Σπόρτερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους αξιότιμους ευρωβουλευτές ε, για τα σχόλια και τις ερωτήσεις και προς τους υπόλοιπους προσκεκλημένους και προς εμένα. Να πω και εγώ κάποια σκέψεις μου ε, σε σχέση με τις μελέτες που έγιναν αλλά και με τα σχόλια που άκουσα. Ε, δεν είναι κάτι το απλό και υπάρχει και ο, ο πειρασμός της υπεραπλούστευσης των ε, πραγμάτων και του κινδύνου και, και πολλής ε, κόσμος ε, πέφτει σε αυτή την παγίδα και ενδίδει σε αυτό το πειρασμό. Κοιτάξτε, η σχέση μεταξύ ε, του κλίματος και της ασφάλειας δεν είναι εύκολη. Νομίζω ότι όλοι το είπαμε και το καταδείξαμε με διαφορετικούς τρόπους. Ε, δεν κάνει κανείς άμεση σύνδεση. Δεν υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού. Αυτό θα ήταν μάλλον αφελές ε, μεταξύ συγκεκριμένων σειράξεων και κλιματικής αλλαγής. Τώρα βέβαια σαφώς υπάρχουν ε, σε πολλές σειράξεις τέτοιες, τέτοιες, τέτοιες συνδέσεις, αλλά εντάξει δεν θα μπω τώρα σε πολλές λεπτομέρειες. Ε, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Βελέρο, ε, κοίταξτε, είπατε για την ανθρώπινη ασφάλεια δεν μιλάμε για τη στρατιωτική έννοια της ασφάλειας. Ε, εντάξει, υπάρχει συχνά μια υπαρξιακή απειλή όταν ε, η γη που μένει κάποιος σταματά να υπάρχει, για παράδειγμα, ή γη την οποία δουλεύει σταματά να υπάρχει. Μιλάμε για πολύ ευρεία ε, έννοια της ασφάλειας όταν διάλεξα τις περιοχές εντάξει δεν διάλεξα το Σαχέλ δεν συμφωνώ ότι το κλίμα δεν έχει καμία σχέση με την αύξηση των πιέσεων εκεί. Ε, το έκανα για να προσπαθήσω να σας ε, δείξω αυτό που θέλω να πω. Ε, δεν μπορούμε βέβαια να υπεραπλουστεύουμε. Η κλιματική διπλωματία τώρα. Εγώ είχα την χαρά του 2000-2001 να ρωτηθώ στην προηγούμενη μου, τότε, στην τότε μου δουλειά, πριν από τέσσερις δουλειές δηλαδή, ε, από τον Επίτροπο Πάτων. Μου ζητήθηκε λοιπόν να εξετάσω την εφαρμογή της διαδικασίας του Κάρντιφ, δηλαδή να συμπεριλάβουμε την περιβαλλοντική πολιτική στι άλλες πολιτικέ και όταν το κάναμε αυτό στι μεταφορές, στις ενέργειες, το να συμπεριλάβουμε λοιπόν το περιβάλλον, όχι το κλίμα, το περιβάλλον τώρα στι εξωτερικέ πολιτικέ, εμπορική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική ε, και τότε την ε, ε, ε, αναδυόμενη ε, ε, κοινή πολιτική, και εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, όταν πριν από ένα χρόνο ανέλαβα τα τωρινά μου καθήκοντα, χάρηκα πολύ που κληρονόμησα ένα λειτουργόν δίκτυο κλιματικής διπλωματίας όχι μόνο στην ΕΕΔ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε, άλλες, σε άλλους τομείς που ε, εργάζονται επί αυτού του θέματος. Ε, εμείς δύο είμαστε που δουλεύουμε στην ΕΙΕΔ για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να είχαμε και περισσότερες, ε, περισσότερες εμπειρογνώμονες, αλλά εν πάση περιπτώσει, στον πραγματικό κόσμο ζούμε. Ε, Ε, συνεργάζονται με το δίκτυο που έχουμε επιτόπου, Του διπλωμάτε μα, τι πρεσβείες τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργαζόμαστε με αυτού του ανθρώπου. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο που μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί με μικρό αριθμό προσωπικού ε, και μιλάω τώρα για το δίκτυο. Τώρα, τα κεφάλαια αηφόρων άπτυξη σε όλες τις ε, συμφωνίες μας. Ε, ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται Επίτροπος Μάλμστρομ να σας το πει αυτό. Μπορώ να σας το πω κι εγώ. Η ιδέα είναι διτή. Θέλουμε να αυξήσουμε τις προδιαγραφές σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω των ε, συμφωνιών ε, με τις οποίες ε, εξεπηρετούμε τα συμφέροντά μας και επίσης προσπαθούμε να επιβάλλουμε αυτή την αύξηση των προδιαγραφών. Αυτό είναι προς συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε, μερικές, σε μερικούς τομείς έχουμε υψηλότερα περιβαλλοντικά, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές, όχι στο κλίμα, αλλά πράγματι με μερικές περιφέρειες του κόσμου, όντως ισχύει. Προσπαθούμε πάντως να υπάρχει μια ισότιμη αντιμετώπιση. Ο ΙΕ. Ναι. Για την αναθεώρηση, την αναμόρφωση του συστήματος του ΟΗΕ, Ε, μιλώ τώρα για τη διατήρηση βέβαια της ειρηνευτικής διάστασης ε, του, του ειρηνευτικού χαρακτήρα του ΟΗΕ και κατά πόσο τώρα έχουμε ηγέτες ε, στην ευρωπαϊκή κλιματική διπλωματία. Έχουμε κάποιες χώρες οι οποίες έχουν κάνει περισσότερα βήματα, έχουν περισσότερο συμπεριλάβει τη διάσταση αυτή στα Υπουργεία Εξωτερικών Μιλήσατε για το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι μόνοι, κάτω χώρες είναι, πρωτοστάτησαν στην ασφάλεια ε, της ε, επάρκειας των ε, φυτών και των καλλιεργειών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και νομίζω ότι κάλυψε το χρόνο μου. Ναι, δυστυχώς είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος μας, λέει η κυρία Φωτίγκα. Ε, γιατί έχουν έρθει ήδη οι ομιλητές μας για το επόμενο πάνελ, για την επόμενη μας ακρόαση. Παρακαλώ να είστε λοιπόν σύντομος κύριε Ρούτιγκερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω ε, σε κάποια από τα σχόλια και στα επιχειρήματα που ακούστηκαν δεν πρέπει να τα αντιπαραβάλλουμε το ένα στο άλλο. Ναι, εντάξει, υπάρχει κάποια πλούστευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, σοβαρές μελέτες ε, δείχνουν όντως ε, ότι το κλίμα και η περιθωριοποίηση είναι πάρα πολύ αποφασιστικοί παράγοντες. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τη σχέση μεταξύ του κλίματος και του ευάλωτου, γιατί θέλουμε να δούμε πώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει το πόσο ευάλωτος είναι κάποιος. Στο Σαχέλ αυτό δεν είναι απολύτως σαφές 100% πώς το κλίμα ε, θα αλλάξει. Οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι θα, υπάρχει, θα υπάρχουν αλλαγές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό, ο αντίκτυπος που θα έχει αυτό έχει να κάνει με την περιθωριοποίηση, έχει να κάνει με το ευάλωτο της περιοχής, Εξαρτάται λοιπόν από αυτούς τους παράγοντες, συνδέονται αυτά τα δύο και δεν θα έπρεπε να ε, θεωρούνται ε, ξεχωριστά ε, το ένα από το άλλο. Είναι ένα επιχείρημα, αυτό ήθελα να πω. Τώρα, όσον αφορά τις λύσεις, γιατί είναι σημαντικό και θα το πω πολλές φορές και πρέπει να το πω πολλές φορές, αν βρούμε λύσεις σε αυτές τις συγκρούσεις και τις σειράξεις, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν πρέπει να αυξήσουμε το πόσο ευάλωτες είναι αυτές οι περιοχές στην κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, όσοι προσπαθείτε να αποφύγετε την περιθωριοποίηση, πρέπει να λάβετε υπόψη την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν παραδείγματα ειρηνευτικών διαδικασιών στην Ανατολική Αφρική, για παράδειγμα, Υπάρχουν ειρηνευτικά κέντρα στις κοινότητες Ανατολικής ε, Αφρικής, όπου μετά γίνεται, υπάρχει ξηρασία. Σε αυτές τις κοινότητες ε, όπου υπάρχουν τα ειρηνευτικά κέντρα, ήταν αυτές πιο ανθεκτικές στην επόμενη ξηρασία, γιατί ήταν καλύτερο το σύστημα διαχείρισης συγκρούσεων και είχαν μια καλύτερη δυνατότητα διαχείρισης των φυσικών πόρων. για παράδειγμα η, κίνηση των, ε, η μετακίνηση των βοσκών που αναφέρατε κι εσείς. Όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν ε, τις προσπάθειες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Δύο ακόμη σημεία και τελειώνω να υπάρχει διαφορετικός αντίκτυπο σε διαφορετικές περιοχές. Είναι σημαντικό αυτό και θα ήθελα να τονίσω και ακούστε και στα παραδείγματα που αναφέρθηκαν σήμερα, να μην βλέπουμε μόνο τι πιο, ε, τις περισσότερο πληγήσει περιοχές όπως το Μάλι και η Συρία, ε, πρόκειται για χώρες οι οποίες ε, θεωρούνταν πιο ανεπτυγμένες, ε, πιο σταθερές και παρόλα αυτά είδατε ότι και αυτές βρίσκονται σε κίνδυνο και αν αυτές οι χώρες κινούνται προς πιο ευάλωτη κατάσταση μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο σε, μπορεί είναι πολύ μεγαλύτερος ο αντίκτυπος από ότι σε χώρες που ήδη είναι ευάλωτες. Και εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με το Υπουργείο Εξωτερικών ε, της Γερμανίας ε, που εδώ και 8 τουλάχιστον χρόνια είναι πάρα πολύ δραστήριο ως προς τον τομέα αυτό. Έχει κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες ε, να συμπεριλάβει αυτό στην ενημέρωση των πρεσβειών να θεωρηθεί δηλαδή η κλιματική διπλωματία μια προτεραιότητα και υποστήριξαν και στο G7 την άποψη αυτή και τώρα προσπαθούν να ενθαρρύνουν στο πλαίσιο ε, του G7 νέες προσπάθειες Και οι κάτω χώρε είναι όλο και πιο δραστήριε για το θέμα τη ε, κλιματική ασφάλεια, αλλά ίσω η Μάλικ να ήθελε να πει περισσότερα προ αυτά. Ο κύριο Μπενιένσεν. Ευχαριστώ. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν αφισβητώ την κλιματική αλλαγή. Το είπα και το ξαναλέω αμφιβάλλω ή αμφισβητώ την ιδέα ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα σειράξεων στην Αφρική. Και αυτό ήταν στην έρευνά μου. Προσπάθησα να αναζητήσω τα αίτια των σειράξεων. Αυτό έχω κάνει. Εγώ λέω ότι αυτή η εστίαση στην κλιματική αλλαγή στις σειράξεις και το Σαχέλ δεν έχει αναφερθεί καθόλου ως περιοχή κλασική σειράξεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Εγώ λοιπόν ανησυχώ ότι αυτή η κλιματική που οδηγεί στη σειράξη του Σαχέλ αποσπά την προσοχή μας από πιο σοβαρά αίτια. Δηλαδή επικαλύπτει αίτια πολύ πιο σημαντικά κατά την άποψή μου. Στο Μάλι δούλεψα πάνω από 30 χρόνια και σπάνια μιλούσε ο κόσμος για κλιματική αλλαγή. Ήμουν στην επίσημη αντιπροσωπεία της νορβηγικής κυβέρνησης το 2008 για την ανάπτυξη. Συναντήθηκα με εκπροσώπους της κοινωνίας, με ηθόντες της κυβέρνησης, οι οποίοι, τους είχαν, είχαν προειδοποιήσει ότι εμένα με ενδιαφέρει κυρίως η κλιματική αλλαγή και είχαμε ενδιαφέρουσες συναντήσεις διήμερες γιατί συζητήσαμε παντού το θέμα της κλιματικής αλλαγής και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια στο Μάλι η πρώτη φορά που άκουσα να γίνεται λόγος για την κλιματική αλλαγή ο κόσμος λοιπόν ανταποκρίνεται θετικά σε αυτά τα αίτια ενδιαφέρεται και τέλος, για τη λίμνη Τσάτ και τη Συρία. Η λίμνη Τσάτ δεν έχει μεταβληθεί σε μέγεθος από την δεκαετία του 70. Συνεχίζει έτσι όπως ήταν. Και αν σας ενδιαφέρει, ο Ζερό Μαγκρέν, καθηγητής γεωγραφίας της γράψε ένα πολύ καλό άρθρο πέρσι με τίτλο περίπου «Ο μύθος της εξαφάνισης Θα το ψάξετε στο Google, θα το βρείτε. Στη Συρία είμαι ένας από τους συντάκτες του περιοδικού «Πολιτική Υγωγραφία» και μιλήσαμε για τη Συρία σε ένα πρόσφατο τεύχος που είναι διαθέσιμο. Μπορεί να σας ενδιαφέρει να το διαβάσετε. Θα ακούσετε λοιπόν και θα βρείτε εκεί όλες τις θέσεις που υπάρχουν σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την σύραξη στη Συρία. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καθηγητά. Η κυρία Μόμπιόρκ. Σύντομα, να σχολιάσω κάποιες ερωτήσεις που ακούστηκαν. Ένας τομέας για, για να χτίσουμε γέφυρες είναι τα κίνητρα. Τα ακούσαμε και από άλλες οργανώσεις. Για να αλλάξουμε τον τρόπο εργασίας μας θα πρέπει να έχουμε κίνητρα. Και η ηγεσία σε μια οργάνωση πώς μπορεί να παράσχει κινήτρα στο να δουλέψουμε διαφορετικά, να αρχίσουμε να ρωτάμε διαφορετικές ερωτήσεις, γιατί για να έχουμε τη δυνατότητα ανταπόκρισης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε μόνο το κίνδυνο αυτό, αλλά έχει να κάνει και με την ε, δικιά μας καθημερινή δουλειά και τον τρόπο που δουλεύουμε. Μπορούμε λοιπόν να ρωτήσουμε τις ερωτήσεις διαφορετικά και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Αυτό είναι το τμήμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και βέβαια ενδεχομένως θα πρέπει να προσθέσουμε πραγματογνωμοσύνη, τεχνογνωσία, αρμοδιότητες κτλ αλλά πρέπει να αλλάξουμε το οργανωτικό μας για να το κάνουμε αυτό. Και έχουμε και ένα θέμα ηγεσία. Εμείς, σε επίπεδο ΟΗΕ, ξέρουμε τι είδο ηγεσία χρειάζεται από πάνω, ώστε οι διάφοροι φορείς μιας οργανωσής να συνεργαστούν καλύτερα σε σχέση ας πούμε και με τη ροή και διάχυση των πληροφοριών μεταξύ οργανώσεων και υπηρεσιών. Και λόγω περιορισμού χρόνου αυτό το παραβλέπουμε. Τέλο πάντων, να τονίσω και να υπογραμμίσω και πάλι το θέμα των κινήτρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Να ευχαριστήσω όλου του συζητητέ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Παρακαλώ, να χειροκροτήσουμε. Thank you very much indeed. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχέδιο γνωμοδότησης είναι το επόμενο σημείο. Θα αφήσουμε να περάσει λίγο χρόνος για να φύγουν και οι συγγητές μας. Ευχαριστώ.

Okay, ladies and gentlemen, please be seated. Λοιπόν, καθίστε παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Our time is limited. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, επαναλαμβάνω. Uh, next point of the agenda, I mean. Ε, θέλω να αρχίσει αμέσως το επόμενο σημείο στη μέση διάταξη. Είναι παρόν ο συντάκτης γνωμοδότησης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Πάσκου. Θα ήθελα εξ ονόματος της ε, Επιτροπής, υποεπιτροπής μας, στο σύνολό της, να σας ε, συγχαρώ ε, για την υψηλή διάκριση που λάβατε πρόσφατα από την Ιαπωνική κυβέρνηση και από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε θερμές ευχές και συγχαρητήρια. Και ας μπούμε τώρα στην ουσία του θέματος που είναι η εξέταση του σχεδίου νομοδότησης ε, βάσει του άρθρου 54 του κανονισμού μας ε, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης με σκοπό τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο πλήρης τίτλος της νομοδότησης. Επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή είναι η Ήτρε και η συγγήτρια εκεί η κυρία Φρανσουάς Γκροστέτ. Uh, uh, και ε, μετά μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, τώρα εξετάζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης και στη συνέχεια Στις 23 το μηνός Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι λίγη προθεσμία για α, την κατάθεση τροπολογιών, οι οποίες τροπολογίες θα συζητήσουμε στο Στρασβούργο. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να συγκαλέσουμε έκτακτη ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας για να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα. Στο Στρασβούργο λοιπόν θα χρειαστεί να γίνει αυτό το Δεκέμβριο, στις 14 Δεκεμβρίου. Τελική έγκριση κάπου το Φλεβάρι, νομίζω. Ενώ προηγουμένως η γνωμοδότησή μας θα έχει εγκριθεί στην ΑΦΕΤ πριν πάει στην Ήτρε. Αυτά. Έχετε το λόγο κύριε Πάσκου για να μην σας καθυστερώ παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια καταρχάς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας γνωρίζετε ε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Είναι πάρα πολύ σφιχτό γιατί είναι πιλωτικό πρόγραμμα διετές και αν δεν μπορέσουμε να το εγκρίνουμε αρχές του 2018 θα χαθεί και δεν θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ για να καλύψει το έτος 2019 και 2020 που είναι η περίοδος για την οποία έχει προγραμματιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζετε ότι γενικά το σχέδιο αυτό έρχεται να συμπληρώσει την ήδη εφιστάμενη παρατηρητικότητα, την ερευνητική, στο ερευνητικό πρόγραμμα, για να καλυφθεί και η φάση της ανάπτυξης, που είναι η πιο ε, έτσι, ρηψοκίνδυνη φάση και πιο δαπανήρη για οποιαδήποτε έρευνα. Καλούμαστε να εφαρμόσουμε. Επίσης, φιλοδοξία είναι να πυροδοτήσει συνεργασία μεταξύ των διαφορών ευρωπαϊκών κρατών. Δεν είναι ε, η πρόθεση να τονωθούν οι εξαγωγές, ούτε ε, προαναγγέλει βαριά στρατιωτικοποίηση, όπως ορισμένοι τείνουν να θεωρούν. Και πιο σημαντικό είναι ότι ενισχύεται τώρα εδώ και αντανακλάται το γεγονός ότι αλλάζουμε υπόδειγμα. Μέχρι τώρα η άμυνα ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και η χρηματοδότηση προερχόταν κυρίως, για να μην πω αποκλειστικά, από τα κράτη-μέλη. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να υποστηρίξει μέσω του περιοδικού αυτού προγράμματος κάποιες φάσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, πράγμα που σημαίνει τι. Ότι ο κρατικός ε, προϋπολογισμός και η κρατική χρηματοδότηση θα εξακολουθούν να είναι εκ των ουκάνευ, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουμε και τη νέα δυνατότητα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο περισσότερα κονδύλια ε, προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τόσο το καλύτερο, τόσο θα αυξηθεί και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να έχει λόγο για, τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανώνται αυτά τα κονδύλια. 30 τροπολογίες περίπου κάναμε για αρχή και μεταξύ αυτών κάτι που λείπει από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε μία σειρά εγγράφων ψηφισμάτων για κατηγορίες όπλων που απαγορεύονται. Αυτά δεν επιτρέπεται να ενταχθούν στο παρόν πρόγραμμα. Εμείς θελήσαμε να βεβαιωθούμε ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και το γράφει η νομοδότησή μας. Γιατί υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την επιλεξιμότητα, διότι από ό,τι φαίνεται η κατάσταση στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από εκείνη που είχαν εκτιμήσει οι συντάκτες και επίσης η πραγματικότητα σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ε, κάποια εξαρτήματα που παράγονται σε τρίτες χώρες. Ε, άρα είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι φανταζόμασταν ή περιμέναμε. Θα πρέπει να βρούμε απαντήσεις σε αυτά και προτιθέμεθα να υποβάλουμε και άλλες τροπολογίες. Και τέλος, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι καλύπτουμε όλες τις σημαντικές και ενδιαφέρουσες πτυχές. Πρώτον, τι κόστος είναι αυτό που θα καλύπτεται, τι είδους είναι το επιλέξιμο, ε, το υπολογιζόμενο κόστος ή το πραγματικό. Ε, άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να διευκρινιστεί. Με ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση του έργου και ποιος είναι ο ρόλος του υφισταμένου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ε, και ποια είναι η δομή που, οι δομές που προτίθεται να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε, διότι ε, αυτό το διαπραγματεύονται τώρα στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη, για να δούμε το αποτέλεσμα των εργασιών. Mm. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε έναν γερό προϋπολογισμό όταν μεταφερθεί αυτό από πιλωτικό πρόγραμμα στην πραγματική ζωή, σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί μέχρι τώρα είπαμε είναι πολιτικό, ε, πιλωτικό πρόγραμμα και τα λεφτά έρχονται από περικοπές άλλων ε, προγραμμάτων. Και θα πρέπει να υπάρξει και κάποια ισορροπία. Διότι κάποια στιγμή κάπου θα πρέπει να ενισχυθούν και άλλες προσπάθειες, όχι μόνο στα οπλικά συστήματα, ας πούμε η προληπτική δημοκρα... Ε, διπλωματία, συγγνώμη, ε, που όλο και περισσότερο αυξάνεται σε σημασία. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια ισορροπημένη χρήση των διαφόρων εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Όπως ε, θα αναμενόταν, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Ορισμένοι μπορεί να πούν ότι δεν φτάνουν τα λεφτά, άλλοι θα πούν ότι είναι πάρα πολλά. Και ξέρετε ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια φάση όπου θα πρέπει ε, σταδιακά να συμπλησιάσουμε τις απόψεις μας για να βρούμε κάποια συνένεση κάπου στη μέση. Οι συνάδελφοι θα κοιτάξουν το έγγραφο αυτό. Θα μας πούν τι θέλουν να προτείνουν ως συνεισφορά και στο Στρασβούργο θα έχουμε όταν πάρουμε όλε τι τροπολογίε την πρώτη συζήτηση με τους και Η πρόεδρος σας είπε το χρονοδιάγραμμα και βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σφιχτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ για τα σχόλια αυτά. Ξέρω ότι είναι παρόντες δύο σκιώδες ηγητές, ο κύριος Δρογεύσκη και η κυρία Βαλέρο και ο κύριος Καστάλτο. There is, uh, uh, any other Άλλος που να έχει εξουδιώτηση να μιλήσει εξ ονόματος και όδους εισηγητού. Εξ ονόματος κύριου Βανόρντεν εσείς, μάλιστα. Ο κύριος Δρογεύσκη αμέσως. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ήθελα καταρχάς ε, να συγχαρώ αλλά και να ευχαριστήσω τον κύριο Πάσκου. Πάρα πολύ καλή δουλειά του. Εμένα με απασχολούσε λίγο να σας πω την αλήθεια αυτή η έκθεση. Νόμιζα ότι θα υπήρχαν πάρα πολλές τροπολογίες που τελικά θα αποδυνάμωναν ε, το νόημα της έκθεσης και την ουσία της. Ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Επίσης, θα, γίνει και, θα υπάρξει και μια γνωμοδότηση της Ήτρε. Ο κύριος Μαρινέσκου είναι υπέρ της ενίσχυσης του Κοπέρνικους και άλλων προγραμμάτων, όπως και άλλες τεχνολογίες ε, και άλλων τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της ε, ε, ε, τεχνολογίας μας στην Ευρώπη. Οπότε εγώ συμφωνώ απολύτως με την άποψη του εισηγητή μας. Πιστεύω ότι θα έπρεπε το παράρτημα να συμπεριλαμβάνει στόχους που δεν θα χρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό θα δείξει ποιες, ποιοι είναι οι στόχοι οι πραγματικοί αυτού του προγράμματος. Επίσης πιστεύω ότι για ένα πιλωτικό πρόγραμμα είναι πολύ σοβαρό εγχείρημα, είναι ακριβό, όπως είπε και ο κύριος Πάσκου, Επίσης, ε, αντλεί χρηματοδότηση και από άλλα προγράμματα. Πρέπει λοιπόν να στεφθεί με επιτυχία όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα εφαρμογής ε, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής προγράμματος, αυτό χρειάζεται περισσότερη προώθηση ώστε να χρησιμοποιηθεί όλο το δυναμικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μην ε, πάει τίποτε χαμένο και να μην ε, αποκλειστούν καλά επιστημονικά κέντρα ούτε χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τις τροπολογίες τώρα του εισηγητή, θεωρώ ότι καθιστούν ε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο ρεαλιστική γιατί επιτρέπουν ε, τη συνεργασία των κοινοπραξιών των κρατών μελών με τρίτες χώρες και γι' αυτό πιστεύω ότι το πρόγραμμα μπορεί να φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι έχουμε μία έκθεση μέσω της οποίας θέλει να ενισχύσει και, το, και την ερευνά της Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κραντσινοντέμσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά που είπε ο κύριος Φανόρντεν που είπε ο συνάδελφο εκ μέρους του κυρίου Φανόρντεν, μάλλον. Ε, εγώ είμαι ε, σκιώδης εισηγητής της ECR στην Ήτρε. Οπότε και εγώ ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο έγγραφο και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την άποψη του κυρίου Στρογεύσκη. Είναι πολύ καλέ οι τροπολογίε του εισηγητή, συμφωνώ σε αυτό. Θα ήθελα όμως να σα επιστήσω την προσοχή σε κάποια θέματα τα οποία τα έθεσε και ο κύριος Πάσκου και ο οποίο πρότεινε μάλιστα και λύσεις. Μιλάω για τις τροπολογίες στις οποίες αναφέρεται ότι αυτές οι αναλογίες πρέπει να εξισορροπηθούν οι διαφορές μεταξύ των ε, παλαιών και των νέων ε, χωρών. Υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια κρόαση σήμερα το πρωί. Σχετικά. Το θέμα δεν είναι μόνο αν πρέπει να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να υπάρχει ένα μεταβατικό πρόγραμμα που θα επιτρέπει ε, τη συμπερίληψη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων από κεντρικές και ανατολικές χώρες Ευρώπης. Σήμερα το πρωί είδαμε το χάρτη που μας παρουσίασε ένας Γερμανός εμπειρογνώμων και ο χάρτης έδειχνε ότι η Βόρειο-Ανατολική Γερμανία Ε, ήταν κρανίου τόπο σε σχέση με τα ερευνητικά ιδρύματα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Το πρόγραμμα αυτό δεν θα έπρεπε να κάνει διπλή δουλειά άλλων προγραμμάτων ε, του ΝΑΤΟ ή πρωτοβουλειών των κρατών μελών. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να είναι συμπληρωματικό και όχι να υποκαθιστά άλλα προγράμματα. Επίσης υπάρχει και το θέμα των ορισμών. Πώς θα ορίσουμε αυτές τις επιλέξιμες ε, ε, εταιρείες, επιλέξιμους φορείς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν ορισμό. Μια ευρωπαϊκή επιχείρηση. Πάρα πολύ στενός είναι αυτός ο ορισμός, γιατί υπάρχουν εταιρείες, οντότητες, οι οποίες συνεργάζονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα με τις Ηνωμένε Πολιτείε, με το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, στο μέλλον. Μια και έχουμε το Brexit. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα είναι τα πράγματα με τη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον. Δεν θα πρέπει πάντως να αποκλείουμε αυτές τις εταιρείε Όμω, οι εταιρείε που θα έπρεπε να αποκλείονται είναι αυτέ που καλύπτονται από κυρώσει ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για τις προσωπικότητες και συμφωνώ με την άποψη που ακούστηκε ήδη στην αίθουσα ότι ήταν πολύ, δεν ήταν καθόλου ξεσορροπημένη η σύνθεση της Επιτροπής, θεωρούμε ότι θα έπρεπε η σύνθεση να είναι πιο αντιπροσωπευτική, να υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα τα κρατημέλη, εφόσον αυτή η Επιτροπή θα τρέξει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί στον αμυντικό τομέα βλέπουμε μεταξύ των κρατών, εντός των κρατών μελών ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και του, του κλάδου. Συμφωνούμε πάντως ε, με εσά, κύριε Σιγητά, και πιστεύω ότι, ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια θαυμάσια εκθέση στο τέλος με τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Βαλέρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πάσκου για το σχέδιο γνωμοδότησης Είναι πολύ ιδιαίτερο λοιπόν το κείμενο το οποίο συζητούμε. 60 χρόνια τώρα ποτέ δεν υποστηρίξαμε την αμυντική βιομηχανία από κονδύλια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Υπάρχει και άρθρο στη συνθήκη που απαγορεύει να χρηματοδοτούμε την αμυντική ε, βιομηχανία. Το έχει παρατραβήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, το πρόγραμμα αυτό που προτείνει μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή, καλούμαστε να υποστηρίξουμε μια βιομηχανία της οποίας το βασικότερο πρόβλημα είναι η υπερπαραγωγή ε, οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη. Επίσης, έχουμε ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία που λόγω αυτής της υπερπαραγωγής της δεν είναι και πάρα πολύ αποτελεσματική. Άρα τώρα τι θα πρέπει να κάνουμε, τους δίνουμε και λεφτά. Στήριξη οικονομική από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Νομίζω ότι έχει σημασία στα διάφορα κράτη-μέλη βεβαίως να υπάρχουν καλές ε, ικανότητες αμυντικές, ε, αλλά αυτή τώρα είναι η ενδεδειγμένη λύση. Εμείς θα καταθέσουμε μία πρόταση μειοψηφία εναλλακτική για την συνεργασία στην έρευνα. Και αυτό που θα προτείνουμε είναι να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία στην έρευνα μεταξύ των κρατών μελών και επίσης σε καμία περίπτωση θεωρούμε δεν θα πρέπει να δοθεί ούτε ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να χρηματοδοτούνται τέτοιου είδους προγράμματα. Και για να επανέλθω ε, στο σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Πάσκου, σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες, ορισμένες από τις τροπολογίες σας. Εδώ αναφέρουμε στην τροπολογία 5 και στην τροπολογία 20, 5 και 20, τα είπε ο ίδιος ο κύριος Πάσκου. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τροπολογία 16, την 29 και την 30. Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να υπάρξει μια σύνδεση ανάμεσα στις δηλώσεις που κάναμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις δράσεις που δεχόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Πάσκο, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, διαφωνούμε και νομίζω δεν θα σας εκπλήξει κάτι τέτοιο. Colleagues, please. Όχι ιδιωτικέ συνομιλίε, λέει η πρόεδρο. Ο κύριο Καστάλτο, παρακαλώ. Ε, <clears throat> thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Πάσκο. Ευχαριστώ, τον ευχαριστώ για τη δουλειά και την προσπάθειά του η γνωμοδότησή του έχει τεράστια σημασία και πάντα παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες αλλά και μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα πάω ντουγρού στο ψητό και θα τονίσω τις ανησυχίες μας αλλά και ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες προτάσεις μας. Καταρχάς θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον κύριο ρόλο τους. Σημαντικό ρόλο για ολόκληρο το βιομηχανικό ιστό της Ευρώπης. Ο ρόλος τους λοιπόν θα πρέπει όχι μόνο να ενισχυθεί, αλλά να προωθηθεί περαιτέρω. Κατά την άποψή μας, ένα τμήμα αυτών των σχεδίων θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά στις μικρομεσαίες και ένα από τα κριτήρια επιλογής αυτών των επιχειρήσεων θα είναι ακριβώς, θα πρέπει να είναι η εμπλοκή δικτύων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διάβασα με ενδιαφέρον τις προτάσεις τροπολογίας σχετικά με τις ε, μικρομεσαίες και την σχέση τους με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Εδώ η απόψη είναι κάπως διαφορετική, γιατί οι μικρομεσαίες κατά την απόψή μας έχουν ε, κάτω από τους 250 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να τις συνδέσουμε με επιχειρήσεις μεγάλες με χιλιάδες εργαζόμενους. Οπότε ίσως θα έπρεπε να αναζητήσουμε μια συμβαστική πρόταση ώστε αυτή να αντανακλά τον ορισμό της μικρομεσαίας. Ένα δεύτερο στοιχείο πάνω στο οποίο θα έπρεπε να παρανεύουμε νομίζω είναι ο ελάχιστος αριθμός, ο απαραίτητος ελάχιστος αριθμός ε, συμμετεχόντων κρατών μελών για να ζητηθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Νομίζω ότι ο αριθμός θα πρέπει να, είναι, να αυξηθεί δηλαδή στο 3, ακριβώς για να διασφαλίσουμε ένα ευρωπαϊκό πνεύμα και το πρόγραμμα αυτό να είναι πραγματικά περιεκτικό και να ξεπεράσουμε ήδη δηλαδή το διμερέ στοιχείο που και αυτό έχει άλλους τρόπους να υλοποιηθεί και να αποφύγουμε βέβαια και το κίνδυνο δημιουργίας ολιγοπολίων και να πάμε προς πολυμερείς και περιεκτικές εμπειρίες. Συμφωνώ αντίθετα την ε, τροπολογία που διαγράφει τι επιχειρήσει οι οποίε κατά 5% ανήκουν σε ευρωπαίου ιδιώκτες. Θα ήθελα να τονίσω και το γεγονό ότι ο έλεγχο τη επιχείρηση πρέπει να είναι σε ευρωπαϊκά χέρια και έχουμε το Golden Share και άλλους μηχανισμούς που αποβλέπουν σε αυτό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να παραβλέψουμε σημαντικές, σημαντικούς μηχανικούς πόρους τη στιγμή που το νομοθετικό πλαίσιο και το βιομηχανικό πλαίσιο μας διασφαλίζει μέσω αυτών των μηχανισμών ότι ο έλεγχος βρίσκεται σε ευρωπαϊκά χέρια. Να επανέλθω τώρα σε κάτι γενικότερο. Τα κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων Εκεί θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα αίτημα για μείωση και απάλληψη των επικαλύψεων υπέρ της βιομηχανίας. Ένας από τους κυρίους στόχους της Ευρωπαϊκής Αμερικής Βιομηχανίας, όχι μόνο για την κάλυψη τεχνολογικών κενών που είναι προφανή, είναι το να δαπανάμε λιγότερο και καλύτερα και θα ήθελα ακριβώς αυτή η προοπτική να ενισχύεται περισσότερο. Τέλος, κάτι πολύ σημαντικό που θα πρέπει να πω για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε το να σταλθούν εσφαλμένα μηνύματα λόγω ακριβώ χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα για χρηματοδοτηθεί αυτό εδώ. Θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τα 40 εκατομμύρια από τη γραμμή του προπολογισμού που αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον και να μην ξεχάσουμε και το Γαλιλαίο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ακριβώς για να αποτρέψουμε παρόμοιες επιλογές γιατί με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα στέλναμε στην κοινή γνώμη ένα πολύ λαθασμένο μήνυμα. Θέλουμε να επωφεληθούμε των ευκαιριών, υπάρχουν σημαντικές ε, προβληματικές, αλλά θα συνεργαστούμε με επικοδομητικό τρόπο για να βελτιώσουμε αυτή την έκθεση, αυτή την γνωμοδότηση. Και να μην ξεχνάμε τις αρχές μας όμως, οι οποίες, ξαναλέω, θα πρέπει να είναι κοινέ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Προσβλέπω στην στενή συνεργασία με εσά και με άλλου συναδέλφου κατά τη διάρκεια τη διαδρομή αυτή τη νομοδότηση. Ευχαριστώ κύριε κύριε Πρόεδρε. Euh, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο Πασκού που συνέταξε μια καλή γνωμοδότηση και συμμερίζομαι ευρέως το περιεχόμενό της. Υπάρχουν δύο σημεία παρά αυτά που θα ήθελα να αφιστώ σε προσοχή σας και να είμαστε πιο προσεκτικοί θα έλεγα. Άξα από κάποιους συναδέλφους κάτι παρόμοιο. Το πρώτο είναι ότι έχουμε να κάνουμε ένα ταμείο άμυνα, το οποίο θα πρέπει να παράγει αποτελέσματα. Αποτελέσματα απτά για τις ένοπλε δυνάμεις μας. Εμείς δεν είμαστε ούτε σε κάτι το καθαρά πειραματικό, ούτε σε κάτι το οποίο αποτελεί ένα νέο ταμείο συνοχής. Δεν είναι ένα διορθωτικό ταμείο αυτό το οποίο είχε δημιουργηθεί για να καλύψει τις καθυστερήσεις των ΜΕ και των ΔΕ σε σχέση με την ε, τεχνολογία άμυνας. Έχουμε να κάνουμε ένα ταμείο το οποίο αποβλέπει στην βελτίωση συγκεκριμένων στοιχείων και ικανοτήτων. Κάποιοι συνάδελφοι το θεωρούν αυτό ως ένα ταμείο που θα καλύψει κενά. Όχι μόνο όσον αφορά το δυναμικό, αλλά και στο βιομηχανικό επίπεδο και σε κάποιες περιοχές συγκεκριμένε. Δεν είναι εθνοτικό ταμείο, έτσι. Να μην το ξεχνάμε, αλλιώς θα ξεχνάμε τι ακριβώς σημαίνει και τι στόχο έχουμε. Δεύτερο σημείο για το οποίο ευχαριστώ την προσοχή σα και κάτι που άκουσα με ανησυχεί ιδιαίτερα γι' αυτό, η ευελιξία για άνοιγμα προ τρίτε χώρες. Εγώ δεν είμαι κατά κάποια μορφή ευελιξία σε σχέση με τρίτε χώρε, μη ευρωπαϊκέ, επειδή βεβαίω σε αυτή τη μηχανία είναι αναπόφευκτο. Βεβαίω, απλά και μόνο δεν είμαι σίγουρο ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει από την αρχή, δηλαδή από την άρξη αυτού του προγράμματος. Αν λοιπόν από την αρχή, από την άρξη του προγράμματος εμείς με μια ευελιξία μεγάλη κάνουμε ένα άνοιγμα σε τρίτες χώρε, οι οποίε δεν το χρειάζονται και τόσο. Να το πούμε ξεκάθαρα, να είμαστε ειλικρινεί. Μιλάω για τι ΗΠΑ, έτσι. Αν η αμυντική βιομηχανία τη Αμερική χρειάζεται ευρωπαϊκά κονδύλια, είναι πιο ε, ανταγωνιστική, είναι αστείο. Να μην λέμε λοιπόν ότι να είναι. Η αμερικανική βιομηχανία είναι παρκώ ισχυρή σήμερα, ήδη για να προσελκύσει τέλο πάντων τα ευρωπαϊκά χρήματα που αγοράζουν αμερικανικά προϊόντα. Δεν χρειάζεται λοιπόν για άλλη μια φορά εμείς να τροφοδοτήσουμε την Αμερικανική βιομηχανία. Δεν έχουμε αυτό το στόχο. Οπότε προσοχή. Γιατί και πάλι υπάρχουν σφάλματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Δεν είμαι κατά της ευελιξίας, είμαι όμως κατά του ευελιξία να αποτελεί ένα μέγιστο απόλυτο κριτήριο από την αρχή. Δηλαδή να απολέπουμε ευθύ εξ αρχής σε αυτό. Εμείς θέλουμε το αντίθετο. Στοχεύουμε στην ευρωπαϊκή και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Καστάλτο και ο κ. Πασκού, ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να οδηγούν ή να αφορούν τον έλεγχο και όχι τους μετόχους, κάτι το οποίο είναι πιο πρόσκαιρο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί αν λοιπόν από την αρχή με τις επιφυλάξεις και τον ευρωπαϊκό προπολογισμό παίρνουμε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογωμένων για να βοηθήσουμε και να ωφελήσουμε τις αμερικανικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις άλλων χωρών, τότε εγώ πολιτικά δεν ξέρω πώς θα μπορέσετε να το στηρίξετε αυτό. Οπότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ευχαριστώ λοιπόν την προσοχή σας σε αυτό. Κατά τα άλλα, θεωρώ το κείμενο του κ. Πάσκου πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει μια πολύ σημαντική βάση για ισχυρές συγκλήσεις. Ευχαριστώ κύριε Ντόνζο. Ο κύριος Λίτς. Ευχαριστώ πολύ στα πολωνικά, κυρία Πρόεδρε. Αγγλικά συνεχίζει ο κύριος Λίτς. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση και τις προσπάθειες που κάνετε. Μιλώ εξ ονόματος των επιτροπών στις οποίες εργάζομαι, το νομικό ζήτημα δεν έχει λυθεί καθόλου. Δεν προβλέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο κάτι τέτοιο. Και χρειάζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ε, εδώ στην υποεπιτροπή υπάρχει μια άποψη στην οποία δεν συμμερίζονται οι άλλες επιτροπές όλες. Ε, υπάρχει πρόταση για εποπτική επιτροπή ε, εν ώψη της έγκρισης ε, εξαγωγών. Συμφωνώ και μου αρέσει αυτό που είπε ο κ. για τις τρίτες χώρες και τη συμμετοχή τους. Δεύτερον, τα θέματα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα και το copyright για προϊόντα που έχουν παραχθεί με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και πιο μακροπρόθεσμα θα πρέπει να κοιτάξουμε από κοινού το μέλλον και η σύγκληση να είναι ε, στο πρόγραμμα. Και τέλος, 125 εκατομμύρια αντί για 500 έχουμε εντάξει στο περιθώριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το παράρτημα για τον ελαφρύ οπλισμό και τη μη εξαγωγή τους. Ε, πολύ σημαντικό βήμα για να προχωρήσουμε. Uh, Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συντομία σας, γιατί είμαστε πάρα πολύ στριμωγμένοι χρονικά. Ο κύριος Στρογεύσκη ήθελε να πάλι και πάλι το λόγο, αλλά πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, ένα λεπτό, ενάμιση θα χρειαστώ σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Ντονζόν, συμφωνώ. Συμφωνώ με την άποψή σας, αλλά θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο εξή. Ο κύριος Πάσκου, στην τροπολογία του που επιτρέπει τις τρίτες, στις τρίτες χώρες να συμμετέχουν, αναφέρει περίφραστα ότι θα δίδεται αυτή η δυνατότητα υπό δύο όρους. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες τεχνολογίες στην Ευρώπη, δηλαδή αν δεν υπάρχει τεχνολογία στην Ευρώπη, αν δεν αντιτίθεται στα ε, συμφέροντα ασφαλείας της Ευρώπης και αν τέτοια συμμετοχή χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα ήδη τρέχον project. Αυτό ήθελα να πω απλώς. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα με τι ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Θα ήθελα να δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Πάσκο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι σημαντικά ε, σημεία, φυσικά θα τα σκεφτώ και μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι θα συνεργαστούμε και περιμένω αγωνία στην πρώτη μας συνάντηση στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και περνούμε ευθύ αμέσω στο επόμενο που είναι ένα εργαστήριο για το μέλλον ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι. Thank you. We start next. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ευθύς αμέσως, το θέμα είναι το μέλλον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Πρόκειται για ένα εργαστήριο και έχουμε εδώ δύο προσκεκλημένους. Ε, δυστυχώς ένας από τους προσκεκλημένους δεν μπόρεσε να έρθει γιατί ασθενεί. Οπότε με πολύ χαρά και τιμή υποδέχομαι τον δόκτορα Κρίστιαν Μόλινγκ που είναι ο αναπληρωτής διευθυντής του ερευνητικού ιδρύματος ε, του Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων ε, και τον δόκτορα, τον καθηγητή Νταβίτ Βερσάγε που είναι ο ε, συνδιευθυντής του νέου ε, ΠΙΚ, δηλαδή των νέων πρακτικών καινοτομίας και δημιουργικότητας στη Σχολή Επιχειρήσεων των Παρισίων Μας ακούει ε, και ο ε, διευθυντής του οργανισμού ε, θέλει να ακούσει τις απόψεις μας για το μέλλον του οργανισμού. Θα ακούσουμε λοιπόν τους δύο προσκεκλημένους και μετά θα ε, δώσω ε, το λόγο σε εσάς στους ε, συναδέλφους. Πρώτος, ο δόκτωρ Κρίστιαν Μέρλινγκ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για τα σχόλιά σας και για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα για αυτό το ενδιαφέρον ζήτημα για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Εγώ δεν μιλώ εκ μέρου τη κυβέρνησή μου. Πρέπει να πω ότι δεν είναι η επίσημη γραμμή της γερμανικής κυβέρνηση της ε, από ό,τι κατάλαβα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Εγώ σας μιλάω με την ιδιότητα κάποιου που δουλεύει στον οργανισμό άμυνας ε, για 10 χρόνια περίπου τώρα ε, με πολλούς ανθρώπους ε, έχω δει τα πάνω και τα κάτω, τις καλές και τις κακές στιγμές ε, του Οργανισμού Αμυνάς. Στις σελίδες που σας έστειλα και στις διαφάνειες προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα όχι θεσμική αλλά του τι θέλουμε να κερδίσουμε από αυτό. Θέλουμε περισσότερη ασφάλεια να βγει από όλη αυτή τη διαδικασία και περισσότερη άμυνα. Και τα ερωτήματα, το θέμα τον, το θεσμικό είναι το δεύτερο ζήτημα που θα καλύψω. Θα αρχίσω λοιπόν τώρα την παρουσίασή μου. Είναι ένα πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, υπάρχει και στο ΝΑΤΟ και ε, σε άλλους οργανισμούς. Υπάρχει ένα πολλά, υπάρχουν πολλά προβλήματα αποτελεσματικότητας προς την άμυνα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Μία τεχνική λύση σημαίνει πολιτικός τετραγωνισμό του κύκλου. Δηλαδή η τεχνική λύση είναι ότι συζητούμε, έχουμε οικονομίες κλίμακας και άλλα πολλά πράγματα που προκύπτουν από τον οικονομικό παράδεισο που μπορούμε να σκεφτούμε. Το πρόβλημα είναι οι κυβερνήσει και ο κλάδος ε, ε, δημιουργούν εμπόδια. Οι κυβερνήσεις γιατί θέλουν να έχουν το δικαίωμα να μπορούν να αποφασίζουν εθνικά. Δεν αναγνωρίζουν παράλληλα ότι δεν είναι θέμα ε, αποφάσεως είναι θέμα δυνατότητας εφαρμογής των αποφάσεων. Η ικανότητα επίλυσης προβλήματος είναι σημαντικότερη από την ε, ικανότητα λήψης αποφάσεων. Θεωρούν όμως, υπάρχει μια ψευδέστηση κυριαρχίας, θεωρούν ότι αν αποφασίζουν θα ε, υπάρξουν αποτελέσματα. Το άλλο είναι ο βιομηχανικός εθνικισμός, ε, δηλαδή η ανάγκη ε, επιστροφής των επενδύσεων στις εθνικές εταιρείες. Αυτό ισχύει όχι μόνο από την, ύπαρξη, από την αρχή ύπαρξης του ε, Οργανισμού Άμυνας, ε, από την αρχή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα αυτό. Το πρόβλημα των κρατών μελών είναι ότι στο τέλος ε, είναι ε, πιο αλληλεξαρτώμενα τα κράτη-μέλη ως προς την εφαρμογή των, αποστα... των αποφάσεων. Κάτι ε, το οποίο βέβαια δεν είναι καλό τώρα. Ο ρόλος και η εξουσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Υπάρχει ένα κενό μεταξύ της, του ρόλου και της, του, πραγματικού του ρόλου και της δυνατότητάς του να δράσει. Και επειδή υπάρχει αυτό το κενό, αυτό το χάσμα, ε, δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει το ακράτη μέλη στον τετραγωνισμό του κύκλου. Έχει μια ισχυρή εντολή από την αρχή που ουσιαστικά ήταν στο πλαίσιο ε, των καλών στιγμών ε, της ε, ΚΕΠΑ τότε Δηλαδή προσπάθησε να δώσει έτσι μία ε, επαναστατική και νέα ε, επνοή ε, σε αυτήν την εξωτερική πολιτική. Όμως ουσιαστικά αυτό εξουδετερώθηκε ε, λόγω της θέσης πολλών εθνικών ε, υπουργείων ε, Άμυνα. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες πίσω από αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εν ολίγης αυτό συνέβη. Η εντολή λοιπόν που είχε ο οργανισμός δεν του επέτρεψε ποτέ να εκπληρώσει την αποστολή του. Για την... Τώρα η συνθήκη της Λισαβόνας πολιτικοποιεί κάπως την όλη διαδικασία, δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων στον οργανισμό για πολιτικά ζητήματα, πολύ πολιτικά πολιτικά ζητήματα ε, για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως σε σχέση με την ικανότητα και τον κλάδο. Ε, το 2007 λοιπόν αρχή της συζήτησης με την εφαρμογή και την, απο... την επιτυχή εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα τότε από ότι τώρα το 2017. Έχει περάσει ο οργανισμός από έναν ε, καινοτόμο οργανισμό σε έναν ε, συντονιστή κατά κάποιο τρόπο λόγω της εξουδετέρωσης του από τα κράτη-μέλη και έχει δημιουργηθεί ένα διαφορετικό τοπίο. Κινούμεθα από μια στιγμή, ε, από μια εποχή κατά την οποία ε, ο στρατιωτικός τομέας ε, έχει πια να κάνει με πάρα πολλούς τομείς πλέον και φορείς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με αυτό το τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Οπότε ουσιαστικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έπρεπε πάντοτε να προσαρμοστεί και δεν ξέρουμε κατά πόσο κατάφερε όντω να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο τοπίο, σε αυτό το νέο περιβάλλον. Ουσιαστικά έχει βυθιστεί στο θεσμικό τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο βέβαια από τη μία είναι καλό γιατί δείχνει μία κανονικότητα, όμως επειδή γίνεται πιο βαρύ το θεσμικό ε, ε, τοπίο, σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες πολιτικές, όμως ο οργανισμός αμυνάς έχει κάπως παραγνωριστεί στο πλαίσιο αυτού του νέου θεσμικού περιβάλλοντος. Τώρα, ε, ποιος θα μπορούσε, ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας είναι ακόμη απαραίτητο, ενδεχομένω και περισσότερο από την παλιά, λόγω των αλλαγών ε, στο περιβάλλον ασφαλεία, ε, στην περιοχή γύρω από την Ευρώπη. Αυτό που θα χρειαζόταν είναι να ενισχυθεί. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι η θεσμική λειτουργία και οι αρχές του να ενισχυθούν, αλλά και μια στρατηγική καθοδήγηση, γιατί για την ώρα υπάρχει μια καταστροφική ε, ασάφεια ε, στην παγκόσμια, στην, στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σλόγγαν που χρησιμοποιεί, δηλαδή πρέπει ο οργανισμός να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης του ΠΕΣΚΟ, του ΚΑΡΤ, του EDF. Ε, υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων μέσων δηλαδή σε σχέση με σε τι βαθμό είναι υποχρεωτικά ή αν μπορεί κανείς να επιλέξει τι θέλει να κάνει και αυτό είναι κάτι ε, στο οποίο δεν μπορεί να, είναι, ε, να διευκολύνει ο οργανισμός άμυνα. Αν το CARD, ας πούμε, παραμείνει ένα εθελοντικό εργαλείο, τότε τα κράτη-μέλη θα εξακολουθήσουν να κάνουν αυτά που κάνουν τα τελευταία δέκα χρόνια, δεν θα δώσουν τα σωστά αριθμητικά στοιχεία, θα αποστηρώσουν όλη αυτή την πληροφορία και ο σχεδιασμό ο που θα γίνει θα βασίζεται σε ένα... Ε, ε, σε μια σαφρή βάση. Ε, η στρατηγική, η αμυντική στρατηγική της Ένωσης, τέλος πάντων η συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτήν, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά και στις διάφορες πρωτεύουσες, δεν είναι αρκετά σαφής. Γιατί μιλάμε, μιλάμε για την άμυνα διαχείριση κρίσεων ή μιλάμε για την άμυνα. Ε, είναι τελείως, διαφορετικό πράγμα. Ε, είναι ακόμα αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αν ε, διαβάσει ε, κανείς αυτά που λέει ε, η πάτη εκπρόσωπος, τότε ε, η άμυνα είναι μόνο διαχείριση της κρίσης. Το ίδιο ισχύει και για τη στρατηγική αυτονομία. Είναι μία από τα, ένα από τα σημαντικά συνθήματα της ε, ε παγκόσμιας στρατηγικής. Αν δει κανείς το επίπεδο της φιλοδοξίας εκεί δεν έχει αλλάξει τίποτε. Δεν έχουν αλλάξει δηλαδή πάρα πολλά πράγματα σημαντικά σε σχέση με τι αποστολέ σε Πέτερσμπουργκ και το επίπεδο φιλοδοξία του 2003. Οπότε τι γίνεται τώρα, υπάρχει κάτι που δεν βλέπουμε στην όλη υπόθεση. Ε, θέλουμε όντω μια προσπάθεια ενίσχυση του οργανισμού Άμυνα ή ε, ε, απλώς πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ασάφεια των όρων που χρησιμοποιούμε. Τι θα πει άμυνα. Αυτό πρέπει να το δούμε και πρέπει να το εξηγήσουμε. Τι είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας αμυνόμαστε έναντι τίνο και τι ποιον θέλουμε να προστατεύσουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ε, ε, σημαντικό και αν δω τη δική μου την πρωτεύουσα ακόμη δεν είναι σαφές. Και τέλο, θα ήθελα να σας παρουσιάσω δύο επιλογές. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες, θα μπορείτε να σκεφτείτε κι εσείς μερικές, αλλά για λόγους αφήνειας δύο επιλογές υπάρχουν. Η μία επιλογή είναι η ενίσχυση που σημαίνει ότι διατηρούμε ε, τη διακυβερνητική διάσταση και ότι είναι μεσολαβητής με τον ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με άλλους φορείς, ε, αυτό έχει την εξή σημασία. Δίνουμε τη δυνατότητα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα να παίζει ένα ρόλο για τι κυβερνήσει και για τα κράτη-μέλη, γιατί ο άμυνα για το προβλεπόμενο μέλλον, εγώ θα στοιχημάτιζα ένα ε, πολύ μεγάλο μπουκάλι σαμπάνια. Θα παραμείνει λοιπόν ένα σημαντικό ζήτημα. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει κάποιο ο οποίο μπορεί να είναι ο μεσολαβητή, ο ενδιάμεσο μεταξύ αυτών που συμβαίνουν στι πρωτεύουσε και καταλαβαίνει τι γίνεται στη φούσκα των Βρυξελών. Να συνδέονται δηλαδή αυτά τα δύο. Τι γίνεται στι Βρυξέλλε με το τι γίνεται στι πρωτεύουσε. Δεύτερη επιλογή είναι να διατηρήσουμε τις λειτουργίες ε, του οργανισμού, να τις ενισχύσουμε, αλλά να ενταχθεί σε ένα ολόκληρο αρχιπέλαγος, ας πούμε, ε, αμυντικού περιβάλλοντος εδώ στην Ευρώπη, να το ενσωματώσουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τον οργανισμό, ε, δηλαδή ακόμη πιο πυκνό θεσμικό μηχανισμό όμως να συνδέεται η άμυνα και η ε, ασφάλεια κάτι το οποίο είναι αυτό που προσπαθεί να πουλήσει ως διαφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον ΝΑΤΟ και άλλους ε, οργανισμούς αμυντικούς. Λοιπόν, από λειτουργική απόψεως αυτό θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Γιατί μέχρι τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προτίθεται να ε, αναλάβει έναν πραγματικό αμυντικό ρόλο κοιτάζοντας πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι θα είχε απολύτως νόημα να συμπεριληφθεί ο αμυντικός πυλώνας ε, σε ένα θεσμικό περιβάλλον ασφαλείας. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αν η απάντηση ε, για τις αλλαγές στην τάξη πραγμάτων που αφορούν την άμυνα είναι απλώς μια αλλαγή ακόμα στην νομική βάση ε, του οργανισμού. Αυτό πραγματικά δεν είναι καθόλου φιλόδοξο και φυσικά, και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, δεν θα παρέχει περισσότερη ασφάλεια. Και τώρα ξαναπάω πίσω σε αυτό που είπα στην αρχή. Εγώ αυτό θα ήθελα να προκύψει από τον οργανισμό, ανεξαρτήτως του ποιο θα είναι το μέλλον του. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνα σήμερα. Θα μιλήσω ως οικονομολόγος. Δέκα χρόνια ήμουν στο Υπουργείο Άμυνα της Γαλλίας. Σήμερα δουλεύω στο Πανεπιστήμιο. Και είμαι πια σε θέση να μιλήσω πιο ελεύθερα. Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω το θέμα των αρμοδιοτήτων στα διάφορα πλαίσια. Όταν συζητάμε αυτό το θέμα, είναι καλό να αναφέρουμε κάποια σενάρια για το μέλλον της υπηρεσίας. Και όταν στην αρχή προετοιμάζαμε την εισηγήση, εξετάσαμε τις διάφορες πτυχές του εγγράφου της Κομισιόν του Ιούνιου φέτος. Το πιο σημαντικό κομμάτι των σενάριων που προβλέπουμε αυτή τη στιγμή εξαφανίζονται λόγω των προσφάτων αποφάσεων από διάφορες υπηρεσίες που αφορούν αυτές τις πτυχές. Εδώ κυρίως έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά στις αρμοδιότητες και τελικά υπάρχει ένα ελέφαντα στο δωμάτιο, όπως λέμε. Όλοι έχουν το ΝΑΤΟ στο μυαλό τους. Αυτό δεν ισχύει, γιατί εδώ ο ελέφαντας είναι το να εισαγάγουμε μια βιομηχανική πολιτική αντί ενός συγκεκριμένου θέματος όπως η δυνατότητα άμυνας. Οπότε να κάνω τρεις παρατηρήσεις εδώ. Η πρώτη αφορά την ανάγκη εστίασης στα θέματα αμυνάς. Η δεύτερη αφορά την εξέλιξη των αρμοδιοτήτων για αυτό τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Και η τρίτη παρατήρηση αφορά άμεσα την διάδραση μεταξύ δραστηριοτήτων προσανατολισμού στρατιωτικού ή πολιτικού. Γιατί εδώ θα πρέπει να προβλέψουμε τη διτή χρήση αυτών των προγραμμάτων. Ένα άλλο κατακτικό σχόλιο. Αυτός ο οργανισμός έχει αναπτυχθεί στο, στα πλαίσια του διοργανικού πλαισίου. Οπότε εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ανάγκη καταγραφής όλων των διακυβερνητικών αλλά αναγκών και μελλοντικών εξελίξεων μεταξύ του διοργανικού πλαισίου και της Κομισιόν. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία. Λόγω ακριβώς της θέσης της είπα της εκπροσώπου και της ύπαρξης αυτού του οργανισμού, εδώ λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να λάβουμε υπόψη μας διάφορα σχήματα διακυβέρνησης ώστε να πετύχουμε συγκεκριμένου στόχους και συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια. Το πρώτο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη δημιουργίας διαφορετικών δυνατοτήτων. Όχι με συγκεκριμένε δραστηριότητε, έρευνας α πούμε ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ βεβαίω υπάρχει ανάγκη διατήρηση του σκεπτικού για θέματα άμυνας επειδή υπάρχει μια μεγάλη σχέση μεταξύ της ε, στιγμής που κάνουμε τη βασική έρευνα στην έρευνα και καινοτομία και της στιγμής όπου θα έχουμε την ε, δυνατότητα να κάνουμε κάτι το οποίο από πλευρά άμυνας θα έχει παγκόσμια κλίση, παγκόσμια έφεση. Εδώ βεβαίως λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε στις δυνατότητες και αυτό είναι μια από τις κυριότητες ε, δυσκολίες σήμερα στο εσωτερικό αυτού του οργανισμού άμυνα. Γιατί όταν συζητάμε αυτές τις πτυχές με άλλους οργανισμούς, με άλλες υπηρεσίε, όταν κάνουμε δηλαδή συγκρίσεις σε εθνικό ή διεθνέ επίπεδο, συνήθως έχουμε τους στρατιωτικούς οι οποίοι συζητούν αυτές τις πτυχές και παρέχουν μια δικιά του σκοπιά. Εδώ θα ήταν καλό να έχουμε ένα μείγμα μεταξύ πολιτών και στρατιωτικών στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Όμως βλέπουμε ότι τελικά κανείς δεν είναι σε θέση να αναπτύξει σταθερή διαδικασία σε σχέση η αιστεία σε σχέση με τις δυνατότητες. Γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού στρατιωτικού. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάγκη για σχεδιασμό και επεξεργασία άμυνας παρόμοια με αυτά που ισχύουν στο ΝΑΤΟ όσον αφορά τα οργανωτικά, την δυνατότητα, το χτίσιμο δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Οπότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό σημαίνει ότι οι αντίστοιχε αρμοδιότητε στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμενα αυτή τη στιγμή, είτε ακριβώ λόγω έλλειψη προσωπικού, είτε ε, λόγω έλλειψη ε, αρμοδιοτήτων δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Επίσης, κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι η ταυτόχρονη εξέλιξη αρμοδιοτήτων και ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Σήμερα υπάρχει μια έλλειψη σύγκληση και μακροχρόνιας κατανόησης μεταξύ των εμπλεκομένων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, επειδή Πράγματι όλοι οι ενδιαφερόμενοι συχνά εστιάζουν σε βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες και θέματα. Και όταν το συζητάμε με όλους, φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό και έχουν ισχυρούς λόγους να το κάνουν. Όταν όμως συζητάμε λεπτομερώς αυτά τα θέματα και όταν παρατηρούμε το πώς κάνουμε αυτή τη δημιουργία δυνατοτήτων σε άλλα περιβάλλοντα, τότε βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει σύγκληση μεταξύ των διαφορών εμπλεκομένων και υπάρχει μια ανάλυση μεθοδολογιών, ανάλυση διαφορών νοοτροπιών εργασίας ώστε να καταλήξουμε σε διάφορες δραστηριότητες και να διοργανώσουμε τις δυνατότητες μας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Θα ήθελα να κάνω τώρα και κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τις αρμοδιότητες Συνήθως όταν συζητάμε αυτό το θέμα από οργανωτική σκοπιά διακρίνουμε σε τρία είδη υπηρεσιών ή οργανισμών. Ένα είδος που θα μπορέσει δηλαδή να αναπτύξει δραστηριότητε παρόμοιες με αυτές που έχουμε στις χώρες όπου Έχουμε δηλαδή τους ε, μηχανικούς ή τελικούς χρήστες στο εσωτερικό των οργανισμών αυτών και μπορούμε να συζητήσουμε ευρέως σε βάθος σε λεπτομέρεια δηλαδή, για τις συγκεκριμένε ανάγκες. Οπότε έχουμε στο εσωτερικό αυτών οργανισμών αρμαδιότητες με αυτές που έχουμε και που αφορούν και τη μηχανία. Βεβαίω αυτό το είδο αρμοδιοτήτων έχει εξαφανιστεί σε όλους τους δημοσίους οργανισμούς παγκοσμίω. Το δεύτερο είδος συνήθως σχετίζεται με τη δυνατότητα διευκόλυνσης δραστηριοτήτων και διάδρασης μεταξύ των εμπλεκομένων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει ακόμα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, θα πρέπει όμως να εστιάζεται με τρόπο πολύ συγκεκριμένο, ώστε να έχουμε επαρκές επίπεδο κατανόησης όσον αφορά τις ε, δυνατότητε από στρατιωτική σκοπιά ή να έχουμε το αντίστοιχο από τεχνολογική σκοπιά, ώστε να βοηθήσουμε τους στρατιωτικούς. Όταν το αναφέρω αυτό, αναφέρομαι και στην ανάγκη κοινή συνεργασίας και δραστηριοτήτων που αφορούν το πεδίο μάχης. Και νομίζω πράγματι ότι η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των εφόρων προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα συνήθως σχεδόν πάντοτε έχει να κάνει με θέματα αντίληψης. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι οποίοι εργάζονται πάντοτε σε θέματα και προγράμματα τεχνικά για την άμυνα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να συζητήσουν ακριβώς με τη βιομηχανία ή με τα συστήματα έρευνας και κοινοτομίας κατά διάρκεια της διαδικασίας που αφορά τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί το να διευκολύνουμε αυτό το είδος ανάπτυξης, το να διευκολύνουμε αυτό το είδος συζήτηση απαιτεί συγκεκριμένε ικανότητες και αρμοδιότητες και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια πρόκληση, γιατί θα πρέπει να το συνδέσουμε με τις διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις. Και άλλη μία επιλογή που αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς όσον αφορά την ανάπτυξη δυνατοτήτων έχει να κάνει με τους οργανισμούς ανάθεσης προμηθειών. Εδώ δεν χρειάζεται να συζητήσουμε με τη βιομηχανία ή του ερευνητέ. Χρειαζόμαστε απλά και μόνο την αρμοδιότητα ή τη δυνατότητα να θεσπίσουμε κάποιε διοικητικέ ε, διαδικασίε, να γίνονται κάποιε συναντήσει κτλ. για να συντάσσονται οι συμβάσει. Αυτό όμω είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που μιλάμε. Γιατί εδώ μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν εσεί δηλαδή εργάζεστε μόνο ω αρχή ανάθεση προμηθειών δεν επηρεάζεται τις ε, συναντήσεις με τον τρόπο που θα έπρεπε ή με τον τρόπο που συνήθως διευκολύνεται την τεχνολογική σκοπιά, τη σκοπιά των επαφών βιομηχανία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα, γιατί όταν αναπτύσσουμε τις εκτιμήσεις μας ε, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, κανείς δεν ξέρει την τοποθεσία, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται ε, με τα επίπεδα δικαιοδοσίας και αρμόδιοτητας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ώστε να είμαστε σε θέση Δηλαδή να μεταφέρουμε τις διάφορες φιλοδοξίες που σχετίζονται ας πούμε, με την ΠΕΣΚΟ, με τα πρόσφατα έγγραφα, με το Ταμείο για την Άμυνα κτλ. Να τα μεταφράσουμε όλα αυτά, να τα ελοποιήσουμε σε συγκεκριμένες δυνατότητες μέσα στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ώστε να τα εφαρμόσουμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι διαφορετικοί κόσμοι που παρουσιάζουν, οι λόγια που παρουσιάζουν τα διάφορα έγγραφα θα παραμείνουν σε επίπεδο ευχολογίων. Οι αρμοδιότητες λοιπόν, ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκάθαρο στο εσωτερικό αυτό των οργανισμών. Και βεβαίω εδώ θα πρέπει να μετατρέψουμε όλες αυτές τις πτυχές σε ένα μείγμα δυσχεριών ή προκλήσεων. Και εμείς όλα αυτά θα πρέπει να τα μετατρέψουμε σε ένα συγκεκριμένο απτό οργανισμό στο πλαίσιο της πικορικότητας διαθέσιμο σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Πώς μπορούμε λοιπόν να μεταμορφώσουμε, να μετατρέψουμε τις αρμοδιότητες τις εθνικές σε ευρωπαϊκές. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτό. Και τα τελευταία χρόνια κανείς δεν το αντιμετώπισε αυτό με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι διάφορες χώρες στο εσωτερικό της ε, Ευρώπης ποτέ δεν εφηγάμισαν τις θέσεις τους. Οπότε εδώ λοιπόν έχουμε μια μεγάλη πρόκληση. Και βεβαίως οι διάφορες χώρες μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τις αρμοδιότητές τους στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία και θα πρέπει οι διάφορες ε, διαδικασίες ευθυγράμμισης να ταυτιστούν μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου. Τώρα βέβαια, ό,τι και να σας πω εγώ εδώ, αναφέρονται σε σημαντικά βέβαια προβλήματα, αλλά το να τα μεταφέρουμε και τα υλοποιήσουμε αυτά στην πράξη είναι τεράστια πρόκληση. Η σχέση τώρα με το ΝΑΤΟ. Η σχέση με το ΝΑΤΟ είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα. Ίσως όμως να μην είναι το πιο δύσκολο να λυθεί. Ίσως επειδή τελικά οι λειτουργικές διαδικασίες εντός στρατιωτικών οργανισμών περίπου θυμεραμίζονται με τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ, οπότε όλες οι σημαντικές χώρες που δαπανούν χρήματα και επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία συμμετέχουν στις ίδιες διαδικασίες του ΝΑΤΟ ταυτόχρονα. Οπότε οι διαδικασίε του ΝΑΤΟ και οι δυνατότητες του ΝΑΤΟ ήδη υπάρχουν στα, στους εθνικούς οργανισμούς των χωρομελών. Εδώ βέβαια υπάρχει ανάγκη διοργάνωσης συγκεκριμένα τη σύγκληση μεταξύ των συμβολών στον ΝΑΤΟ και των συμμετοχών στον ΝΑΤΟ και των συμμετοχών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν έχει και τόσο να κάνει σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά έχει να κάνει σχέση κυρίως με τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο μηχανικών πολιτικών. Επιπλέον εδώ έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη δυσκολία, ότι δεν μπορούμε να δαπανάμε τον ευρώ δύο φορές. Δηλαδή είτε το κάνετε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πραγμάτων, με τις ευρωπαϊκές δυνατότητες ή αλλού. Και θέλω να τονίσω αυτό το αλλού. Αλλά συνήθως, συνήθως Έχουμε δημόσια δαπάνη, η οποία συνδέεται είτε με την έρευνα και την καινοτομία, είτε με τις προμήθειες και επενδύσεις όσον αφορά τις δυνατότητες. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια δυσκολία σύγκληση στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σε διάφορες χώρες, οι διάφορες χώρες της Ευρώπης ε, προτιμούν να δαπανίσουν τα χρήματά τους για δυναμικό το οποίο σχετίζεται με το αμερικανικό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη πρόκληση που δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα, αλλά αντιπροσωπεύει ακριβώ μια μεγάλη δυσκολία που πρέπει να αριθμιστεί σε επίπεδο χωρών μελών. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι η διασύνδεση με τις πολιτικές δραστηριότητες. διαχείριση και δυτή χρήση των τεχνολογιών. Εδώ έχουμε θέματα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και εθνικής διακυβέρνησης, γιατί μεγάλο τμήμα της τεχνολογίας που χρειαζόμαστε ακριβώς για την άμυνα και την ασφάλεια παρουσιάζει πτυχές πολιτικής ασφάλειας, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Όλα αυτά έχουν εκενετής διτή χρήση. Οπότε θα πρέπει να βρούμε τη διάρθρωση μεταξύ, ας πούμε, τα στοιχεία που συνδέονται με το διακυβερνητικό πλαίσιο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και το αφενός και αφετέρου τα διθέσιμα κονδύλια για τους θεσμούς, για τον οργανισμό, τον ευρωπαϊκό και την βιομηχανία για τις πολιτικές δραστηριότητε. Ένα καλό παράδειγμα εδώ είναι μια καλή συζήτηση που γίνεται για το νέο ευρωπαϊκό ουρανό που σχετίζεται ω ζήτημα με διάφορες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, Eurocontrol κτλ. και τη συγκρότηση οργανισμών που δεν ανήκουν πια στο διακυβερνητικό πλαίσιο αλλά υπάγονται στην Κομισιόν και έχουν άμεση σχέση με τη βιομηχανία. Οπότε θα συζητήσουμε πτυχές που έχουν να κάνουν με άμυνα και ασφάλεια, θα πρέπει να έχουμε μια κοινή κρίση μπροστά μας που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, πώς ταυτόχρονα θα έχουμε δυναμικό άμυνας σχετικά ιδιαίτερα με τα κονδύλια για την άμυνα, αλλά και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά να αποφελούμαστε από άλλα κονδύλια, ορίζοντας 2020 ή διάφορα άλλα προγράμματα όπως το ΣΕΖΑΡ. Εδώ έχουμε λοιπόν διάφορους οδικούς χάρτες οι οποίοι δεν συμπίπτουν, δεν συμβαδίζουν. Υπάρχουν διάφορα εθνικά προγράμματα που και αυτά δεν συμβαδίζουν. Έχουμε συγκεκριμένο ζήτημα επειδή τελικά αυτό που θεσπίζουμε αφορούν αυτά που ισχύουν και με το Eurocontrol. Δηλαδή, εδώ είναι απαραίτητο να θεσπίσουμε μια υπηρεσία, μια εμπειρία μάλλον για αυτά τα στοιχεία, για να δούμε πώς θα έχουμε αμυντικό δυναμικό, ώστε να έχουμε ας πούμε, ξέρω εγώ, κοινά αεροσκάφη, ταυτόχρονα κάνοντας πράγματα τα οποία θα εγκυλάγει όλους τους Ευρωπαίους. Αν συγκρίνουμε τα διάφορα κυβερνητικά εθνικά σχέδια, τότε ίσως να είναι πιο έξυπνο να πάρουμε όλες τις πτυχές που αφορούν στατικά και πολιτικά στοιχεία, ώστε να τα συγκεράσουμε και να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Γιατί, να το πούμε ξεκάθαρα, κανείς δεν νοιάζεται από πού προέρχονται τα χρήματα. Σε τελική, μας νοιάζει το να υπάρχει δυναμικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην πράξη. Και αυτό έχει να κάνει και με τη βιομηχανία, δηλαδή τον υπάρχει δυνατότητα για τη βιομηχανία να εκπονήσει μακροπρόθεσμα προγράμματα, χρειάζεται μια λιλουχία προγραμμάτων όπου μπορεί κανείς να μάθει βήμα-βήμα, πρόγραμμα με πρόγραμμα για το πώς ακριβώς θα οργανώνει τις δραστηριότητες του. Και δεν πρέπει εκεί να παρακάμψουμε ενδιάμεσες φάσεις, αλλιώς ε, ακυρώνουμε όλη τη διαδικασία. Θα πρέπει να προασπιστούν και στη βιομηχανία αλλά και στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες αυτές, αυτές οι αρμοδιότητες, να μην χάσουμε λοιπόν το, βηματισμό, το βηματισμό μας και να είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή χρειαζόμαστε δυναμικό το οποίο ε, πρέπει να είναι άμεσα χρήσιμο και αυτό το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση τώρα. Ο κ. Δανζόν ο πρώτος. Δεν ζήτησα το λόγο, λέει ο κ. Δανζόν. Δεν θέλετε. Όχι. Καλά. Παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βαλέριο Μπριάνη λέγομαι, εργάζομαι για, ε, στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να απαντήσω στα όσα είπαν τα μέλη του πάνελ. Είναι πολύ χρήσιμη πρωτοβουλία μετά το σάλο που έχει γίνει στην αμυντική κοινότητα. Συμφωνώ ότι ε, ο οργανισμός μέχρι τώρα ε, υπό χρησιμοποιείται, το έχει αναγνωρίσει αυτό η παγκόσμια ε, στρατηγική. Αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς αδρανούμε ότι είμαστε άεργοι. Υπάρχουν τα προγράμματα ε, που συνεχίζονται μέχρι τώρα για 430 εκατομμύρια για το σχηματισμό ικανοτήτων ε, για ένα οργανισμό που έχει 30 εκατομμύρια προπολογισμό και 140 υπαλλήλου δεν είναι και άσχημα. Και αυτό καλύπτει όλο το φάσμα έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη, ε, κατάρτιση, εκπαίδευση, συντήρηση και προμήθειες. Δημόσιες προμήθειες ε, ουσιαστικά. Για τη δημιουργία ικανοτήτων, επαναλαμβάνω. Και επίσης έχουμε και μια σειρά ε, δραστηριοτήτων που δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήματα υποστήριξη μικρομεσών επιχειρήσεων, διασυνοριακή συνεργασία. Αναφερθήκατε στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Εκεί ακριβώς είναι το φόρουμ που έρχεται η στρατιωτική κοινότητα για να συζητήσει. Και εργαζόμαστε για την τυποποίηση, για την πιστοποίηση. Έχουμε ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και θεμάτων που μας απασχολεί. Τον περασμένο Μάιο οι Υπουργοί Άμυνας ενέκριναν το τελικό φάκελο ε, μετά από μία διαδικασία υψηλού επίπεδου συναντήσεων ενός έτους για τη μακροχρόνια αναθεώρηση με τρεις προτεραιότητες να ξεχωρίζουν για τον οργανισμό μας, για το μέλλον. Πρώτη προτεραιότητα και συνδέεται αυτό με τα προηγούμενα που είπατε, είναι ότι θα πρέπει να δρά ως βασικό εργαλείο ε, ιεράρχησης προτεραιοτήτων διακυβερνητικών. Δηλαδή υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη να καταλάβουν τι λείπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον, όχι σε εθνικό, έτσι ώστε να μπορούν να ε, τα καλύψουν πλήρως ή εν μέρη με συνεργασίες. Έχουμε τα νέα μέσα λοιπόν εντάσσονται εδώ όπως είναι το CARD, ε, μια ατζέντα για την έρευνα ε, και κομβικές στρατηγικές δραστηριότητες. Αυτά για τη χάραξη προτεραιοτήτων. Και βέβαια το σχέδιο δημιουργίας ικανοτήτων είναι ένα σχέδιο το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να καταλάβουμε τι χρειάζονται τα κράτη βράχη, μέσο και μακροπρόθεσμα. Δηλαδή συνεργαζόμαστε και με εκείνους. Και Στη συνέχεια, η δεύτερη προτεραιότητα θα είναι να συνεργαζόμαστε. Σας ανέφερα τα 400 εκατομμύρια και προσθέτουμε και νέα προγράμματα, νέα έργα, ε, ας για τον κυβερνοχώρο ή την κινητικότητα τη στρατιωτική. Και επίσης διευκολύνουμε, είμαστε διευκολυτέ δηλαδή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους οργανισμούς και κεντρικός ε, διαχειριστή των ερευνητικών δραστηριοτήτων με κοινοτική χρηματοδότηση. Δηλαδή θα είμαστε ένα είδος σύνδεσμος ε, διευκόλυνση των σχέσεων των κρατών μελών και των στρατιωτικών με του οργανισμού Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. υποστηρίζουμε δραστηριότητες όπως είναι το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Έχουμε ιδιαίτερο ρόλο στο ε, πιλωτικό πρόγραμμα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που συνδέονται ε, με την πτέρυγα της άμυνας, της αμυντικής έρευνας μάλλον. Και προβλέπεται να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια με την υποστήριξη των κρατών μελών για να έχουμε καθαριστικό πρωταγωνιστικό ρόλο και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Άμυνα. Επίση για τις αρμοδιότητες και το προσωπικό θα ήθελα να επανέλθω. Πάνω από τους μισούς υπαλλήλου είναι στρατιωτικοί. Και όλοι οι project officers που εργάζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη ικανοτήτων στα, ε, στις ομάδες εργασίας με τα κράτη-μέλη είναι στρατιωτικοί Ζητώ συγγνώμη, υπάρχουν βουλευτέ που θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Και τελειώνω. Ευχαριστώ. Κύριε Ντανζό. Ε, Καλά. Ε, ε, δεν είναι από υπερβολική τύπο λατρεία. αλλά είμαι εδώ δύο θητείες και για πρώτη φορά βλέπω συζήτηση να γίνεται εδώ με διαφορετικό τρόπο και να διοργανώνεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι είναι με τους ε, προσκεκλημένους και τους ε, βουλευτές. Ε, έχω όλο το σεβασμό για τον εκπρόσωπο του οργανισμού είτε είναι μέλος του πάνελ και θα περιμέναμε να είναι μέλος του πάνελ είτε είναι ακροατής. Το λόγο δεν μπορεί να πάρει κάποιος έτσι διαδικαστικό. Δεν θα πρέπει να είναι ένα τέτοιο προηγούμενο που να επαναληφθεί. Καλούμε κόσμο, τον ακούμε και συζητάμε βουλευτές. Αν μετά ο καθένα πρέπει να έρχεται εδώ και να δικαιολογεί την ύπαρξή του, χαθήκαμε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που δεν είχα ε, προγραμματίσει. Ε, ζητώ συγγνώμη γιατί θα είμαι πάρα πολύ ε, έτσι ρεαλιστικός και, και, ε, Αυτά που μας είπατε είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ θεωρητικά και πολύ λυρικά. Αλλά αυτά που ακούσαμε τώρα ε, έχουν να κάνουν με όλο το μύθο γύρω από τον ε, προορισμό, την αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας κτλ. Γιατί παρόλες τις ε, εξηγήσει που ακούμε δεν είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα και οι θέσεις. Πολιτικά μιλώντας, ένα από τα... Όσα είπε ο Κρίστιαν Μέλινγκ έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα παραμείνει διακυβερνητικός οργανισμός, του οποίου ε, το ισχυρό ατού είναι ο διακυβερνητικό χαρακτήρας, γιατί ξέρουμε ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ έντονο στα αμυντικά θέματα, το διακυβερνητικό στοιχείο. Ή μήπως θα ενταχθεί κάπου, θα εσωματωθεί, embedded το είπατε στα αγγλικά, ε, ε, σε μια αρχιτεκτονική που τώρα δημιουργείται. Πώς να πω, θα είναι ένας πάροχος υπηρεσιών δηλαδή. σε μια υπηρεσία που αναπόφευκτα θα εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ αλλάζουμε λοιπόν τρόπο διαχείρισης ε, για να μην αλλάξουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Χθε συναντήθηκα με τον κύριο Ντομέκ και ε, το ξέρω ότι μπορεί να φανεί και ερετική ερώτησή μου αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βάλει το χέρι στην τσέπη και βαθιά. Οπότε τι θα γίνει, μηχανικά το κοινοβούλιο θα αναλάβει ένα ρόλο αυξανόμενο ως προς τον έλεγχο των ε, διαδικασιών αυτών και των δράσεων. Ακούω όλα αυτά που λέγονται για τον απολογισμό του οργανισμού άμυνας. Δεν φταίει ο ίδιος ο οργανισμός, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και εκτιφλωτικός. Και θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω την άποψή σας γι' αυτό. Δεν έχω αποκρισταλωμένη άποψη εγώ, ούτε για τον οργανισμό τον ίδιο, ε, αλλά πώς βλέπετε τις εξελίξεις, προς ποια κατεύθυνση το πάμε, ποιο είναι το πιθανότερο. Γιατί αν είμαι σίγουρος για κάτι, το, το status quo δεν μπορεί να διατηρηθεί έτσι για πολύ καιρό γιατί πολιτικά εγώ δεν φαντάζομαι τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν σαν να μην τρέχει τίποτα ε, για να διαιωνίζεται μία δομή η οποία δεν πρόκειται να έχει πολύ συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα βράχη πρόθεσμα. Ευχαριστώ. Thank you. Just to respond. Ευχαριστώ για να απαντήσω στις ε, παρατηρήσεις σας. Είναι λίγο δύσκολο από πλευρά μου να ενθαρρύνω του βουλευτέ να πάρουν το λόγο. Σε γενικέ γραμμέ προσπαθώ, αλλά προσπαθώ να μην το κάνω. Ε, Μόλι βλέπω ότι κάποιο θέλει από του ευρωβουλευτέ να πάρει το λόγο, προσπαθώ να σταματήσω τι ε, άλλε παρεμβάσει εξωτερικών. Προφανώ έχουν προτεραιότητα οι ευρωβουλευτέ. Δεν, δεν έχουν αλλάξει οι κανόνε προ αυτό. Απλώ ε, δεν υπήρχαν ε, δεν υπήρχαν ευρωβουλευτές που να έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν ε, τώρα να σας ζητήσω να πάρετε το λόγο, πρώτα ο Δόκτωρ Μέρλινγκ και μετά ο καθηγητής Βερσάγια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό που είπε ο Αγνοντόζο. Η... Εσείς κοιτάτε την πολιτική πλευρά δεν μπήκα στις λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο λέτε δείχνει ότι ακριβώς πρέπει να υπάρχει μια πολιτική απόφαση για το μέλλον γιατί η δομή δεν πρόκειται να αλλάξει επειδή υπάρχει μια εξέλιξη στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Βλέπουμε εδώ μια χαρακτηριστική ένδειξη αυτού που εμείς ως πολιτικοί αναλυτές βλέπουμε ως ζητήματα επιβίωσης. Ε, φαντάζομαι ότι συμφωνούμε ως προς την προοπτική Νομίζω ότι ε, πράγματι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να φέρει αποτελέσματα ο οργανισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 430 εκατομμύρια. Ε, η χώρα μου έχει, έχει 33 δις τζίρο από τα ε, αμυντικά και από τα και από τα άλλα προϊόντα 270 δις. Λοιπόν, αν θέλει λοιπόν να υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος ε, μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα, τότε πρέπει να οριμάσει αυτός ο οργανισμός, είτε οργανισμός άμυνας είτε κάτι άλλο. Ε, πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το έχουμε κάνει κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Αν θέλετε να μπείτε στη δομή προϋπολογισμού της διακυβερνητική χρηματοδότητας του ενός του άλλου πράγματο, στι καλέ στιγμέ ε, τη ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνα, ήταν τέλος πάντων μια γκρίζα ζώνη. Ε, δεν θα έλεγα ότι ήταν κάτι εκτός νόμου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και απολύτως διαφανές και αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε. Γιατί υπάρχουν και οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι που θα δώσουν λεφτά. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα χρήματα θα δαπανώνται με το σωστό τρόπο και για το σωστό σκοπό. Και για μένα τουλάχιστον ως Ευρωπαίο φορολογούμενο έχει σημασία, δεν έχει σημασία κατά πώς λέγεται ο οργανισμός, αρκεί να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό στον τίτλο, γιατί ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά χρήματα είναι αυτά που ξοδεύονται. Λοιπόν, τώρα, το τι μπορεί να κάνει ο οργανισμός, να το πω διαφορετικά, το καθήκον που έχει, γιατί υπάρχει τεράστιο ιστορικό υπουργών άμυνα που εξηγούν πόση εμπιστοσύνη έχουν στον οργανισμό, ε, ναι, ε, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε γίνει από το 2013. Αν δει κανείς το τι έχει ε, ε παραγάγει ως προϊόν ο οργανισμός, αυτό ακριβώς είναι που θα έπρεπε να σκεφτόμαστε για να καθορίσουμε το μέλλον. Γιατί υπήρχε μία έρευνα το 2015, έδειξε ότι δεν φταίει ο οργανισμός, φταίει αυτά είναι τα κράτη-μέλη που είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την ε, πορεία του. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Ε, υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ συντηρητική προσέγγιση αυτή. Θέλουμε να συνεχίσει, θέλουμε να είναι ένας πολιτικός οργανισμός που ε, αυτή ήταν και η ιδέα όταν ιδρύθηκε ο οργανισμός. Αν πάει κανείς πίσω στη σύμβαση ε, στο κεφάλαιο 7 που οδήγησε στη συνθήκη στη συντελεκτική συνέλευση το κεφάλαιο 7 της οποίας οδήγησε στη συνθήκη στη, στη, Λισαβόνα ε, πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ε, πραγματικά ε, παλεύει για την επιβίωσή του οργανισμός ε, και το καταλαβαίνω. Δεν είναι μόνο όμως θέμα επιβίωσης του οργανισμού αυτού, είναι θέμα επιβίωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, νομίζω ότι τα, ε, ο ρόλος των κρατών μελών πρέπει λίγο να ε, τεθεί εν αμφιβόλο. Εφόσον κάνατε την ερώτηση στα γαλλικά, θα σας απαντήσω στα γαλλικά. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Κρίστιαν Μόλινγκ, όμως θα ήθελα να προσθέσω κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, χωρίς να αμφισβητήσω καθόλου το οποίο, αυτό που παρουσιάστηκε ως απολογισμός. Πράγματι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στα αποτελέσματα της δραστηριότητες ε, και ε, των ε, μέσων του περιβάλλοντος, τέλο πάντων μεταξύ όλων των υπολείπων και του στόχου βέβαια που έχουν τεθεί. Η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω για να σας απαντήσω είναι πολύ απλή. Για όλες αυτές τις εργασίες που έχουμε κάνει, ε, όταν βλέπαμε ας πούμε, το θέμα της εξέλιξης ε, των οργανισμών, ε, διακυβερνητικών ή όχι, δεν έχει σημασία. Πολύ συχνά βρισκόμαστε ενώπιν μιας κατάστασης όπου το καθήκον του οργανισμού διαμορφώνεται όχι ε, σκεπτόμενοι ε, την, ε, ε, τα αποτέλεσμα, το τι θέλουμε να επιτύχουμε, αλλά μία ας πούμε πολύ ε, θεωρητική κατάσταση των πραγμάτων, θεωρητική θεώρηση των πραγμάτων. αν δείχνουμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία είναι εντελώς στρεβλή, διαμαρφώσαμε ε, το καθήκον βάσει των αρμοδιοτήτων και όχι βάσει των στόχων. Πρέπει να κάνουμε το αντίστροφο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι που θα επιτύχει τους στόχους των διαφόρων εγγράφων που υπήρξαν για την ΠΕΣΚΟ και για ε, πολλά άλλα ε, προγράμματα. Λοιπόν, για το δεύτερο ερώτημά σας, κοιτάξτε, να το δούμε λίγο διαφορετικά αν υπάρχει ε, ένας οργανισμός που έχει έναν ενδιάμεσο μεσολαβητικό ρόλο, ε, η βασική ικανότητα θα είναι, ας πούμε, κάπως ουδέτερη, θα μπορεί ουσιαστικά να δημιουργεί ε, διάλογο για να μπορέσει να υπάρξει συνένεση, να κινηθούμε προς ένα στόχο. Αλλά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ρόλο, ας πούμε, έμπιστου, ε, πρέπει να υπάρξει μια εικονότητα και πρέπει να υπάρχουν ικανότητες και σε επίπεδο εξοπλισμού και σε επίπεδο ε, ε, τεχνολογικό. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Προφανώ υπάρχουν ε, στρατιωτικέ ε, στρατιωτική ικανότητα στο πλαίσιο του οργανισμού. Αν δει κανεί το προφίλ των στρατιωτών, στρατιωτικών που πρέπει να δουλέψουν στι διάφορε αποστολέ στα κράτη-μέλη ή, στο, ή ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, ε, βλέπουμε ότι ε, είναι τελείω διαφορετικό αυτό από τα αρχικά καθήκοντα για τα οποία είχε δημιουργηθεί ο οργανισμό άμυνα. Αν δούμε, α πούμε, τι γίνεται ε, στη Γαλλία και στη Γερμανία, Γερμανία ε, δεν ε, υπερβαίνουν οι υπεύθυνοι ποτέ το ε, βαθμό του, του συνταγματάρχη. είναι... Είναι πολύ ανώτεροι λοιπόν οι βαθμοί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Ε, γιατί τα κράτη-μέλη ε, στέλνουν σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό και ε, οι άνθρωποι αυτοί μετά διακόπτουν τις σχέσεις τους με το εθνικό επίπεδο. Όμως πρέπει να γίνεται το αντίθετο. Πρέπει να είναι πιο καλές αυτές οι σχέσεις για να υπάρχει ένας πραγματικός προβληματισμός, για να υπάρξει καλύτερη συνένεση μεταξύ των ικανοτήτων που πρέπει να υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο και αυτών που θα δημιουργηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα αυτό που συμβαίνει εδώ και αυτό που βλέπουμε με την ε, βάση της εμπειρίας μας είναι μια αδιάφορη σχέση. Δεν είναι αυτό που μας χρειάζεται όμως. Και καταλήγω στο ερώτημα που θέσατε, αν θέλουμε να σκεφτούμε το διακυβερνητικό, ε, είναι κάτι ε, το οποίο πολλές φορές δεν θέλουμε να θυσιάσουμε καθόλου ανεξαρτήτως του τι θέλουμε να επιτύχουμε. Αυτό το διακυβερνητικό κομμάτι είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα στο πλαίσιο του οργανισμού άμυνας. Δεν πρέπει να το θυσιάσουμε. Τώρα κατά πόσο είναι αρκετό, μάλλον όχι. Και θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπα στο τέλος παρουσίασης μου. Τόσα πολλά πράγματα σήμερα έχουμε να κάνουμε από κοινού με ε, τις ε, ε, τεχνολογίες της διτής, διπλής χρήσης που δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο σε επίπεδο κυβερνητικό. Οπότε θα πρέπει να ξεφύγουμε και από αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει να συμπληρώσουμε τους μηχανισμούς, όχι να είναι η κατάσταση του ενός από του άλλου, γιατί θα έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να ενθαρρύνουμε τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των μηχανισμών. Και για να σας απαντήσω, ποτέ δεν πρέπει να θυσιάσουμε το διακυβερνητικό κομμάτι, απλώς να το συμπληρώσουμε. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια ευκαιρία την οποία μπορούμε να αξιοπιστήσουμε, γιατί... Ε, η σημερινή ε, εκπρόσωπος Είπα ότι εκπρόσωπος ούτως ή άλλως ε, έχει μία καλή ε, στάση ως προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τις τρεις προκλήσεις που πρέπει να αναλάβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τους συγητές μας και όλους σας που συμμετείχατε σε αυτό το workshop. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί έχουμε τη συνεδρίασή μας που αρχίζει 9 Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.